Buenos días. Take seat, please. favor, vamos a... Καλώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε ή καλύτερα να συνεχίσουμε θα έλεγα τις συνεδρίες της Επιτροπής μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους μαθητές τεσσάρων εκπαιδευτικών κέντρων αλληλείας της οποίου τους οποίους έχουμε ανάμεσά μας εδώ. Τους ε, συγχαίρουμε για τις επιλογές τους, τους καλωσορίζουμε. γιατί εργάζονται και σπουδάζουν έναν τομέα τον οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, τον οποίο υπερασπιζόμεθα φανατικά και είμαστε σίγουροι ότι προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Προσπαθούμε να είμαστε οι αντιπρόσωποι σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους για μια ακόμη φορά. Η κυρία Τομά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το καλωσόρισμα των λεγόμενων ναυτικών λυκείων της Βρετάνης. Ε, οι μαθητές αυτοί ασχολούνται με την αλληλεία ή με τις υδατοκαλλιέργειες γενικότερα. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι οι συνάδελφοι α, μερικές φορές αμφιβάλλουν για το κατά πόσον ενδιαφέρουν τα επαγγέλματα αυτά τους νέους. Παρόλα αυτά Υπάρχουν νέοι οι οποίοι, ε, τους οποίους προσελκύει η θάλασσα και ό,τι σημαίνει η θάλασσα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους μαθητές αυτούς των λυκείων της Βρετάνης να έλθουν εδώ και να γνωρίζουν πού λαμβάνονται οι αποφάσεις οι οποίες θα τους επηρεάσουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Σας ευχαριστώ κυρία Τομά. Όπως είχαμε συνεννοηθεί. Περνάμε στο 9 της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τον Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό και τις παρεκκλήσεις από τον ενισχύει κανονισμό. Έχει το λόγο ο κύριος Αρσένης. Παρουσιάζουμε σήμερα την ε, έκθεση για ένα είδος αλίας που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο αντικείμενο. Όχι μόνο γιατί μιλάμε για ψάρια τα οποία διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά που ψαρεύουν οι ψάράδες μας συνήθως. Αυτά ε. που συζητάμε σε αυτή την Επιτροπή. Όχι μόνο γιατί μιλάμε για ψάρια τα οποία ε, ζουν σε πάρα πολύ ακραίες συνθήκες αλλά και γιατί είναι ελάχιστοι ψαράδες στην ε, Ευρώπη που έχουν σαν αντικείμενο αλίας τους αυτό το είδος ψαριών. Μιλάμε για μια πάρα πολύ ειδική κατηγορία. Ψάρια τα οποία ζουν στα άκρα βάθη των ε, ωκεανών μας. Το, για τη σημαίνει περιοχή που συζητάμε είναι η τεράστια αυτή περιοχή του βόρειο-ανατολικού, Ατλαντικού ψάρια τα οποία ζουν σε συνθήκες πλοίους ε, σκοταδιού στην πράξη υπό συνθήκες πίεσης με πάρα πολύ χαμηλό μεταβολισμό που τι σημαίνει σημαίνει ότι έχουν πάρα πολύ χαμηλό ρυθμό αναπαραγωγής έχουν, ε, ε, ζουν πολλές φορές ως και τα 100-150 χρόνια ενώ φτάνουν στη ηλικία αναπαραγωγής πολλές φορές μετά τα 35 τους. Αν σκεφτούμε ε, τι σημαίνει οι νότιες χώρες ε, Πολλέ φορέ παραπονιούμαστε στην Νότια Ευρώπη ότι τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι μετά τα 30 του. Ε, αυτά είναι ψάρια τα οποία φτάνουν σε ηλικία αναπαραγωγή στα 35 χρόνια μερικέ φορέ. Επίση είναι πάρα πολύ άσχημα ψάρια. Ψάρια που για να τα πουλήσουμε στο εμπόριο θα χρειαστεί κάθε φορά ε, να κόψουμε το κεφάλι, να τα κόψουμε σε φιλέτα και να τα προσφέρουμε σαν λευκό ψάρι στους ε, καταναλωτές. Αυτά τα ψάρια δεν τα ψαρεύαμε στην πράξη, δεν, δεν προσπαθούσαμε να τα ψαρεύσουμε στην πράξη. Γιατί ήταν πολύ βαθιά για να φτάσουμε. Ξεκίνησε η προσπάθεια αλλία όταν κατά τη δεκαετία, μετά τη δεκαετία του 60-70 και μέσα το 80 η κατάρρευση των ελιευμάτων στην, ε, στις θάλασσες μας, στις παράκτης περιοχές μας, οδήγησε τους ψαράδες μας να αναζητήσουν άλλα είδη αλληλείας. Γι' αυτό και έγινε αυτή η προσπάθεια να, να μετακινηθούν προς τα βάθη των ωκεανών που κανείς δεν ήθελε να πάει γιατί προφανώς κοστίζει πάρα πάρα πολύ να, στις, σε βενζίνες και σε όλο το, τα καύσιμα που χρειάζονται για να φτάσει κανείς σε αυτές τις περιοχές και να ψαρέψει. Έτσι ξεκίνησε αυτή η αλία και έχουμε... Όμως, επειδή ακριβώς αυτά τα ψάρια ζουν σε τόσο ε, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η μικρή και παραμικρή και πόσο μάλλον μια μεγαλύτερη πίεση στους πληθυσμούς τους οδηγούν σε κατάρρευση. Έτσι τι είχαμε. Το πιο κλασικό παράδειγμα που γνωρίζουμε στην Ιλλανδία το Orange Raffi. Το 2000 στην ουσία ξεκινάει η αλία αυτού του είδους ε, και με επιδοτήσεις και με ενίσχυση από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Το 2002 έχουμε την κορύφωση της, ε, των ε, ε, ψαριών, δηλαδή την έχουμε τα περισσότερα κάτσεις, ε, γίνεται πλέον μια επικερδής αλληλευτική δραστηριότητα και μάλιστα ε, το, η καινούργια εναλλακτική στα ψάρια της παράκτητας περιοχής που ε, έχουν μειωθεί σημαντικά και όμως μέχρι το 2005 μόλις σε πέντε χρόνια έχουμε την κατάρρευση του είδους. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι όλη αυτή η αλληλευτική ευκαιρία καταστρέφεται. Και το 2005 έως σήμερα, το 2013, 8 χρόνια, έχουμε μηδέν επιτρεπόμενη ε, αλία. Έχουμε μηδενικό τάκ. Και δεν γνωρίζουμε πότε θα αποτεσταθεί αυτό το είδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέτρα για την αντιμετώπιση, για την ρύθμιση της αλίας ε, των, αυτών των ειδών βαθιά θάλασσα, το deep sea fisheries. Όμως έχει αποδειχθεί ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν. Έχει αποδειχθεί ότι τα ίδια αυτά δεν αποκαθίστανται. Με ελάχιστε εξαιρέσεις που υπήρξε τα, πέρυσι μια μικρή βελτίωση στα τάξη, τα τάξη κατά, κανόνα ε, είναι χαμηλά, ε, μηδενικά και τα ήδη αυτά δεν μας δίνουν μεγάλες ελπίδες αποκατάστασης. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε με μια πρόταση η οποία λέει δεν θα προτείνει να μην απαγορευτεί η αλληλεία αυτών των ψαριών αλλά να απαγορευτούν να σταδιακά να, να μειωθούν και, και τελικά να απογορευτούν μέσα από ένα, μιας phase-out ε, στρατηγικής τα εργαλεία που προκαλούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ποια είναι αυτά. Έχουμε τα σειρώμενα εργαλεία βυθού, τα bottom sea trawlers, τα οποία γνωρίζουμε από τις, ε, από τις, από τις επιστημονικές μελέτες που παρουσιάστηκαν και εδώ στην Επιτροπή μας ότι προκαλούν παρεπτύπτουσα αλληλεία στα επίπεδα των 144 με 144 148 ειδών όταν οι, οι αλληλείς μας που στοχεύουν τα ψάρια των βαθέων υδάτων στοχεύουν πολύ λίγα είδη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση της Επιτροπής αφορά τη συνέχιση της αλληλευτικής αυτής δραστηριότητα με την αποφυγή των επιπτώσεων ενός εργαλείου που για το συγκεκριμένο είδος αλίας είναι μη, μη επιλεκτικό. Στην, επίσης υπάρχει το phasing out των, των gillnets. Την ίδια Άρα η πρώτη επιτροπή αφορά το να, μεταφερθούμε, από την ε, αλία μέσω ε, των ε, deep sea trawlers στα long lines, στην πράξη τα παραγάδια. Τι σημαίνει αυτό, όπως δήλωσαν και οι επιστήμονες που παρουσιάστηκαν στο, στην ακροματική ε, διαδικασία, αλλά και η Επίτροπος Δαμανάκη από την επίσκεψή της στις Αζόρες, στο κέντρο της βαθιάς θάλασσας της Ευρώπης. Ε, μία χρονιά αλληλείας με bottom sea trawlers ισοδυναμεί στις επιπτώσεις για τα ψάρια βαθιάς θάλασσας σαν 800 χρόνια αλίας με long liners. Αυτή είναι η τρομακτική σχέση. Η Επιτροπή επίσης προτείνει το πάγωμα της αλληλευτικής δραστηριότητας, της, του, του του αλληλευτικού. Τι σημαίνει αυτό. Άμα, επειδή όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, οι ψαράδες μας ε, έχουν το VMS και δίνουν σήμα για το πού ψαρεύουν, πού βρίσκονται κάθε στιγμή στη θάλασσα, κάθε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ξέρουμε αυτό το αποτύπωμα της, ε, του κάθε ε, ψαρά και η πρόταση της Επιτροπής είναι σε αυτές τις περιοχές όπου ψάρευαν να συνεχίσουν να ψαρεύουν και αν χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές να υπάρχει πρώτα ένα, μια εκτίμηση επιπτώσεων, ένα impact assessment ε, για να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Μιλήσαμε για τα ψάρια βαθιών υδάτων. Δεν μιλήσαμε για κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η περιοχές αυτές, ο βορειοανατολικός Ατλαντικός, είναι ο χώρος ενός δύο άλλων πολύ σημαντικών ειδών που είμαστε υποχρεωμένοι διεθνώς να προστατεύσουμε. Είναι η... τα κοράγια, κοράγια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι πιο παλιά από την ιστορία της δικιάς μου χώρας της Ελλάδας και είναι και τα σφουγγάρια, τα σπάντζις. Και τα δύο αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ως είδη και προσφέρουν πάρα πολλές υπηρεσίες σε όλους μας ε, με τον καθαρισμό των νερών και πάρα πολλά άλλα ακόμα. Όμως προσφέρουν μια σημαντική υπηρεσία στο αντικείμενο που ερχόμαστε να συζητήσουμε εδώ πέρα. Και το αντικείμενο αυτό είναι η ανάκαμψη των ειδών των ψαριών βαθιάς θάλασσας. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι ακριβώς τα κοράγια και όπως ξέρετε για τους ε, υφάλους και τις κοραγίνες υφάλους τα κοράγια στο βυθό της θάλασσας και τα σφουγγάρια είναι οι χώροι όπου θα προστατευτούν τα μικρότερα ψάρια μέχρι να μεγαλώσουν, μέχρι να μπορέσουν να φτάσουν μια ηλικία που θέλουμε εμείς για την, για την αποκατάστασή τους της αναπαραγωγής. Γι' αυτό και στην πρότασή μου, όπως θα δείτε, υιοθέτησα την πρόταση συναδέλφων εδώ πέρα στην Επιτροπή για την χωρική προστασία των ευαίσθητων αυτών περιοχών, των vulnerable marine ecosystems, των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, του, της θαλάσσιων οικοσυστημάτων, που είναι τα κοράγια και τα σφουγγάρια. Η πρόταση είναι το ΆΙΣΕΣ, το επιστημονικό όργανο που συμβουλευόμαστε εδώ πέρα στην Επιτροπή ε, αλίας πολλές φορές για την επιστημονική μας δουλειά, ιδίω για αυτή την περιοχή της Ευρώπης, που έχει στοιχεία ε, και έχει πλέον μέσα από τις μελέτες που μας παρουσιάστηκαν και εδώ πέρα στην Επιτροπή, ε, μοντελοποιήσει το πού είναι πιθανό να υπάρχουν τέτοια, τέτοιες περιοχές, τέτοια ευαίσθητα οικοσυστήματα κοραϊών και σουγαριών που είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε, να προτείνει αυτές, να ορίσει αυτές τις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει ε, αλία ε, βυθού ε, και σε αυτές τις περιοχές που βέβαια όμως εφόσον το κράτος μέλος κάνει νες, κάποια νέα επιστημονική έρευνα και δείξει ότι τελικά η περιοχή ήταν διαφορετικά, έπρεπε να υπάρξει διαφορετική χάρη στην περιοχή ή δεν υπήρχε καν αυτή η κρίση, αυτά τα, τα είδη στην περιοχή. Υπήρξε κάποιο Λάθο ή υπήρξε ήδη καταστροφή της περιοχής και δεν υπάρχουν πλέον. Ή εφόσον το, το κράτος εγγυηθεί ότι βάλει τα μέτρα προστασία ώστε να υπάρχει η εγγύηση ότι η αλληλεία σε εκείνη την περιοχή δεν θα πειράξει ε, τους, τα κρίσιμα αυτά οικοσυστήματα, μπορεί ξανά να ανοίξει η περιοχή σε αυτή την, ε, η αλληλεία σε εκείνη την περιοχή. Επίσης, ακολουθώντας την πρόταση ε, άλλων αλλιέων της, ε, ε, του Ατλαντικού ε, αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος που έχουμε εδώ πέρα και την εισηγήτρια την κυρία Άννα Ρόσμπαχ που είναι και σκιώδη εισηγήτρια από το ECR στην έκθεση αυτή και μόλις χθε ψηφίστηκε η έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με 58 ψήφους υπέρ και μία ε, κατά ε, διακομματικά και προτείνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος να υπάρχει ένα, ένα, limita ένα death limitation, ένας περιορισμός βάθους στην αλία αυτής της περιοχής στα 200 μέτρα. Η δικιά μας πρόταση είναι τα 400 μέτρα και είναι τα 400 μέτρα γιατί αυτή είναι η ορισμός του Deep Sea Fisheries από την Επιτροπή στην έκθεσή της, όπου θα δείτε ότι αναφέρει η Επιτροπή ότι θα πρέπει να καταγράφονται με ειδικό τρόπο οτιδήποτε, οποιοδήποτε ψάρι πιάνεται κάτω από 400 μέτρα. Ε, για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό το μέτρο. Ξέρουμε ότι ήδη όπως το Orange Rafi, αλλά και το Blue Link που έχουμε, ε, για τα οποία έχουμε μιλήσει πριν έχουν την τάση να μαζεύονται σε κοπάδια περισσότερο από τα συνήθη ψάρια. Έχουν αυτό το aggregative behavior. Ψαρεύοντας ε, σε, χαμηλότερο βάθη, αυξάνει τον κίνδυνο να πιάσουμε ολόκληρα κοπάδια, ολόκληρα schools ψαριών. Επίσης, με τον death limitation προστατεύουμε ε, πλήρως πλέον τα, τα nesting grounds, τα spawning grounds, όλα αυτά τα, τις περιοχές που είναι τόσο σημαντικά για την αναπαραγωγή των ψαριών που θέλουμε να αποκατασταθούν. Βέβαια, όπως έχω πει σε πολλούς συναδέλφους, ο ορισμός του βάθους ε, αυτού είναι θέμα συζήτησης με το εξής κριτήριο. Οι προτάσεις που υπάρχουν σε αυτή την ε, έκθεση και που καταθέτω εγώ στην Επιτροπή είναι προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν σε έναν στόχο, την προστασία την, ε, των ε, ευαίσθητων οικοσυστημάτων που αναφέραμε και έχουμε την υποχρέωση να τα προστατεύσουμε συμβατικά και διεθνώς, τα σφουγγάρια και τα κοράγια και την αποκατάσταση των ε, ειδών αλίας βαθιάς, των, των ψαριών βαθιάς θάλασσας, δίψη φύσης Δεν αποσκοπεί να έχουμε παράλληλες επιπτώσεις σε άλλα είδη ψαρέματος. Αν, παραδείγματο χάρη, υπάρχει κάποιο είδος, ε, είδη, είδη αλίας τα οποία, ε, αν η απαγόρευση αλίας κάτω από 400 μέτρα οδηγεί σε οικονομική, σημαντική οικονομική ε, ζημιά γιατί ακριβώς ε, είναι, υπάρχουν στοιχεία ε, ότι η πλειονότητα των κάποιο άλλο είδους ψαριού ψαρεύεται χαμηλότερα από αυτό το βάθος προφανώς είμαστε εδώ πέρα να το συζητήσουμε. Η, ο σκοπός της πρώτης αυτής δεν είναι να, να αγγίξουμε άλλα είδη αλληλείας. Και γι' αυτό μάλιστα θα δείτε ότι από την πρόταση, η πρόταση μου ως εισηγητής είναι το Κοινοβούλιο να ζητήσει την εξαίρεση από τη λίστα των ψαριών βαθιάς θάλασσας δύο ειδών, του Kangaroo και του Link, γιατί με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν είναι είδη τα οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να είναι στη λίστα των ψαριών βαθιάς αλίας για, ακριβώς ακολουθώντας αυτή τη λογική. Η πρόταση αυτή που καταθέτω στην Επιτροπή για συζήτηση είναι μια πρόταση για την προστασία ε, την αποκατάσταση των ε, ειδών βαθιάς θάλασσας χωρίς παράλληλες ε, επιπτώσεις, χωρίς ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα, στις άλλες αλληλευτικές δραστηριότητες Έχουμε μια εξαιρετική ακραία περίπτωση ψαριών ειδών θαλάσσιας ζωής παίρνουμε σπάνια μέτρα τα οποία δεν δημιουργούν κανένα είδος προηγούμενο ακριβώς για την αντιμετώπιση αυτής της εξαίρεσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέλω όμως να κλείσω επισημάντως ότι αυτή η πρόταση που καταθέτω στην Επιτροπή για συζήτηση θεωρώ ότι είναι και περιβαλλοντικά, αλλά και κοινωνικά κυρίως και οικονομικά βιώσιμη. Περιβαλλοντικά το έχω εξηγήσει, δεν χρειάζεται να το περισσότερο. Οικονομικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά το κόστος για τα καύσιμα στο οποίο οδηγεί η χρήση των bottom seat rollers σε αυτά τα βάθη της θάλασσας αλλά και σε αυτές τις αποστάσεις τόσο μακριά από ε, τις, τις ακτές μας. Η πρόταση να, να, να μετακινηθούμε στα long lines σημαίνει πολύ λιγότερο κόστος σε καύσιμο. Σημαίνει λιγότερο κόστος στους Ευρωπαίους ε, φορολογούμενους αλλά και λιγότερο κόστος και στα κράτη-μέλη. Όμως και κοινωνικά. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η μετάβαση στα long lines σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας. Ένα κόστος όμως φέρνει όφελος στην απασχόληση. Το δε αυξανόμενο κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με την εξοικονόμηση από τα καύσιμα. Οπότε πραγματικά για το συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης, των αλλιέων μας και της θαλάσσιας ζωής από την οποία εξαρτώμαστε, πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σένη. Έχουμε 7 ευρωβουλευτές που ζήτησαν τον λόγο με την κυρία Τόμα. 8. Το λέω για να ξέρουμε ποιο χρόνο έχουμε. Εσείς Γκαρσία Γέρο, κυρία, έχετε και εσείς ζητήσει να παρέμβετε. 9. Έχουμε λοιπόν μέχρι και, τε, και τέταρτο και 20 πάνω κάτω χρόνο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε με την ελευθερία που δίνουμε στις παρεμβάσεις, αλλά το δυνατόν συντομότερο για να παρέμουν οι περισσότεροι. Ο κύριος Γκάλαγκερ. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον συνάδελφό μας. Εκτιμώ την ε, πρότασή, σου, την πρότασή του να δεσμευτεί ως προς, προς αυτό το θέμα της ε, βαθιάς αλίας για μένα το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους αλείς του Ατλαντικού και είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τον βασικό κανονισμό. Και ανησυχώ ιδιαίτερα με αυτά που άκουσα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος εχθές ότι έγινε μια ψηφοφορία ε, εχθές και από τα 600 μέτρα να κατεβούν στα δύο. Όχι σε τέσσερα, στα δύο. Εάν αυτό λοιπόν είναι το μέλλον, θα υπάρχουν ψάρια, αλλά δεν θα υπάρχουν αλλοίς. Τα 200 μέτρα είναι ένας αριθμός που δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία κατανόηση για το πώς ε, δουλεύει ο τομέας. Και ιδιαίτερα επικροτώ τους 7 συναδέλφους από την Άλντε, οι οποίοι καταψήφισαν τα 200 μέτρα η, τα ψάρια αυτά είναι ένας θησαυρό ε, για μας. Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες, πρέπει να εξασφαλίσουμε την επιβίωση τους για μελλοντικές γενιές. Αλλά δεν πρέπει να ε, καταλήξει όλη αυτή η προσπάθεια στο να καταργηθεί η αλληλεία στο μέλλον. Έχουμε και αυτή την ευθύνη. Όπως ε, Είπαμε νωρίτερα σήμερα, κάθε δάσος ε, δεν είναι και παρθένο δάσος. Λοιπόν, κάθε... Δεν είναι ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο του βυθού έχει κοράλια και ένα βυθό γεμάτο κοράλια. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις του ωκεάνιου βυθού που είναι αμμώδης, ε, έχει φύκια. Άρα λοιπόν ε, δεν πρέπει, δεν έχουμε κανένα λόγο να ζημιώσουμε τα, τις εκτάσεις αυτές που έχουν ε, σπόγγους και κοράλια ε, και χρειάζονται την απόλυτη προστασία μας. Πρέπει λοιπόν η εκμετάλλευση αυτή των ψαριών αυτών να γίνει με, με σεβασμό και έχοντας υπόψη πάντα μια αηφόρο αλία που να μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ας κοιτάξουμε την ε, σημερινή κατάσταση. Αν δούμε τι συμβαίνει σήμερα, ε, ε, επιβάλλονται μέτρα. Μέτρα ισχύουν για να προστατεύσουν το ευάλωτο θαλάσσιο σύστημα όπως κοράλια και σπόγκους τις περιοχές αυτές. Είναι ευάλωτες ε, διότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στο θαλάσσιο περιβάλλον εκεί και πρέπει να το προστατέψουμε. Λοιπόν, η αλία βαθαίου ύδατος, βαθαίων υδάτων απαγορεύεται ήδη στις περιοχές αυτές και μιλάμε για εκτάσεις 12.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Και εάν επεκταθούμε περισσότερο, προτείνουν άλλα 30-35 ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα ως προστατευμένη ζώνη. Όλη αυτή η περιοχή λοιπόν εκτός ε, των υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάμε για 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα οποία είναι ε, κλειστά. Η περιοχή αυτή είναι κλειστή. Απαγορεύεται δηλαδή η αλληλεία εκεί. Άρα λοιπόν δεν είναι ε, αμεληταία, αμεληταίες αυτές οι προστατευόμενες εκτάσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, ε, επιβάλλουμε <clears throat> να υλοποιήσουμε, εφαρμόσουμε πρόσθετα μέτρα ε, βάσει της γραμμής που παρουσιάζει η Κομισιόν στο έγγραφό της. Ε, πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας μία ισόρροπη και ανάλογη προσέγγιση, την αρχή της αναλογικότητας δηλαδή και την δυνατότητα εκμετάλλευση των διεθνών υδάτων. Θα πρέπει λοιπόν τα μέτρα αυτά να επεκταθούν περαιτέρω από τα διεθνή υδατά στα ευρωπαϊκά υδατά. Και αναφερόμενος στα διεθνή ύδατα, ε, με εξαίρεση τις προτετευόμενες εκτάσεις, οι αλληλείς έχουν την υποχρέωση να ε, αποσύρουν τα δίχτυα τους όταν εισέρχονται ή πλησιάζουν, είναι στα όρια των προστατευόμενων περιοχών, να τα αποσύρουν, να τα σηκώσουν, να τα μαζέψουν και να πάνε αλλού. Ε, τα μέτρα που θέλουμε να εφαρμοστούν πρέπει να είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα και ομοιόμορφα, να εφαρμόζουν ομοιόμορφα στα ευρωπαϊκά υδατά. Ε, γι' αυτό ε, προτείνεται λοιπόν η αλία με παραγάδια θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Ισχύει όμως αυτό. Η αλή με ε, παραγάδια θα οδηγήσει στην αλληλεία ε, creating uh, further problems. And... παράπλευρων αλλιευμάτων, ε, ιδίω στην αλληλεία βασαίων υδάτων. Και όπως είπαμε, τα ψάρια που ζουν σε αυτά τα βαθιά νερά είναι βάλωτα. Και ενδέχεται η αλληλεία με παραγάδια να έχει καταστροφικό αποτέλεσμα σε άλλα αποθέματα, σε άλλα αλλιευτικά αποθέματα. Εάν λοιπόν ε, αλλάξουμε από μεσικές στράτες σε παραγάδια μπορεί, χωρίς να το θέλουμε, να καταστρέψουμε παραδείγματο χάρη την αλία της γλώσσας και άλλων ψαριών, αθέλητα. Η Κομισιόν λοιπόν και αυτό με απογοητεύει Ιδιαίτερα πρότεινε 600 μέτρα, συνάδελφοι πρότειναν 400 μέτρα και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, πρότεινε 200 μέτρα. Έχει πάει κανείς να δει πώς γίνεται η αλληλεία στην ε, νοτιοδυτική περιοχή της Ιρλανδίας, όπου βασικά ψαρεύονται γαρίδες. Όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως γαρίδες. Εάν λοιπόν αλλάξει η αλία από τράτε σε παραγάδι, αυτό σημαίνει ότι θα πεθάνει αυτή η αλία της γαρίδας στην περιοχή μας. Δεν είναι λοιπόν μόνο το θέμα της αλίας των ειδών ε, που ζουν στα βασιά ύδατα. Θέλουμε να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ αυτών που θέλουν την πλήρη απαγόρευση και αυτών που θέλουν να επιτύχουν ένα συμβιβασμό. Ο στόχος μας είναι κοινός και πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο με αυτή τη συζήτηση και με την ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με συνεργασία να καταλήξουμε στον κοινό στόχο. Εγώ ξέρω την κατάσταση, είμαι ενημερωμένο. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στην υπεραλίευση του Orange Raffin, δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η υπεραλίευση. Είναι μια κακή κατάσταση. Το orange ruffin ήταν ένα ψάρι το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά έχει τελείως, τελείως ε, ε, πλέον ε, το αλλιευτικό απόθεμα αυτού του είδους. Τελείωσε. δεν υπάρχει πια στην αρχή υπήρχε η αλία του Orange Raffin, γινόταν κανονικά, μετά άρχισε να μειώνεται το απόθεμα, υπευλήθηκαν ποσοστώσεις και τελικά εξαφανίστηκε το είδος. Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν και αντιφάσεις στην πρόταση της Κομισιόν. Στο άρθρο 1 λέει ο στόχος είναι να εφαρμοστούν τεχνικά μέτρα στη διαχείριση της αλίας στο βορειο ε, Ατλαντικό. Το κείμενο όμως δεν αναφέρει παρακάτω ένα συγκεκριμένο μέτρο, όπως λέει ας πούμε στο άρθρο 1. Και η Κομισιόν απέτυχε στο να διαβουλευθεί το STCF και όλες ε, τις συναφείς, όλους τους ενδιαφερόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλίας βασέων υδάτων. Δεν ε, διαβουλεύτηκε. Και ο βασικός κανονισμός συστήνει ή λέει, ορίζει ότι θα πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Και εν καταλήξει θα σας αναφέρω τις πρόσφατες πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσα στα πλαίσια ε, της χρηματοδότησης της βασιάς αλίας. Η Κομισιόν εξέφρασε τις απόψεις της τον Ιούλιο, ξέροντας ότι η έκθεση αυτή θα εκδοθεί τέλος του χρόνου. Και εν κατακλείδη η τελευταία μου λέξη είναι να κάνουμε περισσότερες διαβουλεύσεις, περισσότερες περισσότερο διάλογο και συζήτηση για να μην ε, εξαφανίσουμε και σκοτώσουμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για το παράδειγμα αυτό που δεν είναι καλό από πλευρά χρόνου, από πλευρά σα ή από πλευρά μου που σα άφησα να μιλήσετε, τέλο πάντων να μην συνεχίσουμε. Έτσι έχετε τον λόγο εσεί παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Κρήτον Αρσένη για όλο το έργο που επετέλεσε για αυτό το θέμα και για τον φιλικό συναδελφικό τρόπο που μας προσέγγισε και ήταν πρόθυμος να έρθει να μας τα εξηγήσει. Αλλά θέλω να προσθέσω την φωνή μου σε αυτά που μόλις είπε ο Πατ Δεκόπ Γκάλαχαρ. Διαρωτώ με σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υποβάλλεται μια παρόμοια πρόταση, όταν προτείνεται απόλυτη απαγόρευση της βαθιάς αλληλεία και αν αντικατασταθεί με τα παραγαδιάρικα, ποια τεκμήρια και έρευνα έχουν γίνει σε σχέση με όλα αυτά. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο εισηγητής να μου απαντήσουν το εξής ερώτημα. Πόσα σκάφη στη Σκοτία είναι αυτά τα οποία θα αποσυρθούν από τη δραστηριότητά τους με την επιβολή αυτού του μέτρου σε σχέση με παράδειγμα αυτά τα οποία ψηφίστηκαν εχθές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ΕΝΒΗ 200 μέτρα δηλαδή ως όριο όταν λέτε εσείς ο ίδιος κύριε Αρσένη ότι ο ορισμός ε, της ε, αλίας, βαθιάς αλίας είναι 400 μέτρα και χθε υπερψήφισαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Ένβη του Ευρωκοινοβουλίου 200 μέτρα. Έχουμε στα 900 μέτρα αλία από τους Σκοτσέζους αλίες ε, και εσείς τι προτείνετε τώρα να ξαναγυρίσουμε σε μια κατάσταση και να πούμε στους ε, αλληλείς μας ότι πρέπει να χρησιμοποιούν παραγάδια για να αλλιεύουν αυτά τα αλλιεύματα. Αυτό δεν γίνεται. Θα μείνουν άνεργοι στα λιμάνια. Είναι παράλογη αυτή η πρόταση. Γελία και παράλογη. Και το λέω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πάτε πρώτα να μιλήσετε με αυτούς τους ψαράδες δεν καταστρέφουν αυτοί τους ε, υφάλους, ε, ούτε πλησιάζουν καν τα, ε, τους υφάλους, διότι καταστρέφουν τους γρίπους τους, τα δίχτυα τους. Και έτσι λοιπόν παραμένουν κοντά στην υφαλοκρηπίδα, Porcupine Μπάνκ για παράδειγμα σε σχέση και με τις περιοχές αυτές αλίας και πιο κοντά και στα νησιά Σέτλαντ, ε, παρότι εκεί είναι πολύ ψυχρά τα νερά και πολύ λίγα ψάρια μπορούν να επιβιώσουν. Στην άλλη όμως τάφρο ψαρεύουν μέχρι 900 μέτρα βάθος. Αν απαγορεύσουμε αυτό και σου πούμε δεν επιτρέπεται παρά μόνο παραγαδιάρικα να έχετε μέχρι 200 μέτρα τέρμα η αλία. Κατεβάζουμε τα ρολά και θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με το πρόγραμμα το οποίο δείχνουν κιόλα και στην ε, τηλεόραση την καταστροφή που υπάρχει με γρήπους ε, στα Ριχάνερα Και εκεί ακριβώς ε, εκεί θα καταλήξουμε. Πρώτα θα απαγορεύσουμε τη βαθιά λία και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε με απαγόρευση της, ε, των γρήπων παντού, οπουδήποτε. Και η μεγαλύτερη δραστηριότητα αλληλείας ε, για τις ε, γαρίδες δηλαδή θα καταστραφεί στη δική μας περιφέρεια. Και δεν είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Δεν, καταστρέφουμε ούτε σε σχέση με τα αλλιεύματα, ούτε τους υφάλους βαθέων υδάτων. Πρέπει να έρθουν επιστήμονες να τεκμηριώσουν με επιχειρήματα όλα αυτά και αν εσείς εμένετε και επιμένετε να επιβληθεί αυτή η πρόταση, πού θα πάνε όλα αυτά τα σκάφη που θα αποσυρθούν από αυτές τις δραστηριότητες. Θα πάνε ήδη σε περιοχές που υπεραλλιεύονται και με την εντατική αλληλεία είτε θα υπάρξει καταστροφή αλλιευμάτων είτε καταστροφή Τη της δραστηριότητας ε, στην αλληλεία. Έχουν μόνο αυτή τη δυνατότητα οι δικοί μα αλληλεί. Είναι πολύ εύκολο όταν μιλάει κανεί για τη Βαλτική ή τη Μεσόγειο, όπου δεν έχουμε αυτού του είδου τις ε, ε, βαθιές, βαθέων υδάτων πελαγικές αλληλείας να λέμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο όριο. Αλλά Πιστέψτε με, είναι απόλυτα ανέφικτο να γίνεται αυτό στις περιοχές που εκπροσωπώ εγώ ως πολιτικός. Σας ευχαριστώ η κυρία Ρόντος, που είναι, ε, ε, Ρόσμπακ που είναι η συγγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω δανέζικα. Θα υπάρχει μετάφραση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα ήθελα να με χαρακτηρίσετε σαν το φρικιό της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Δεν είναι αυτή η θέση μου και δεν είναι αυτή η δουλειά μου, αλλά ακόμα και από την δική μου πολιτική ομάδα φοβάμαι ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί βουλευτές να πούνε ότι ας απορρίψουμε ό,τι πιάνουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Δεν πρέπει ξαφνικά να χάνουμε τα αλλιεύματα έτσι όπως συμβαίνει τώρα. Τώρα, για την αλληλεία στα μεγάλα βάθη είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και δυστυχώς μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ε, θα διαπιστώσουμε δυστυχώς ότι ε, οι ηχθειοπληθυσμοί σε μεγάλα βάθη δεν είναι σε θέση να επιβιώσουν. Όπως είπε ο συνάδελφος Αρσένης, είναι, ε, για, πρόκειται για είδη ψαριών τα οποία για να φτάσουν στην φάση της αναπαραγωγής έχουν ανάγκη από το πέρασμα πολλών δεκαετιών. Δεν μπορούμε λοιπόν με τη λογική αυτή να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εξοπλισμούς οι οποίοι μας βοηθούν ακόμα και σε πολύ μεγάλα βάθη να βρίσκουμε τα ψάρια αυτά και να τα αλλιεύουμε. Η λογική αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πράγματι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος υιοθετήθηκε η γνωμοδότηση με 50 τόσες ψήφους υπέρ και μόνο μία κατά. Και νομίζω ότι αυτό κάτι δείχνει. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία στο σύνολο των πολιτικών ομάδων. Ε, για τα 200 μέτρα αν δεν κάνω λάθος αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές ε, δεν ξεπερνούν τα 100 μέτρα, αλλά παρόλα αυτά ε, γνωρίζουμε ότι τα 400 μέτρα είναι το διεθνές επίπεδο το οποίο ε, γίνεται αποδεκτό. Στην ίδια την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, είπαμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση προς όφελος όχι των αλλιέων είναι αλήθεια αλλά των ιδίων των αλλιευμάτων. Διότι οι αλλιείς θα παραμείνουν αλλιείς εφόσον υπάρχουν αλλιεύματα. Αλλιώς τι συζητάμε. Πρέπει λοιπόν να μην περιορίσουμε το ενδιαφέρον μας στους αλληλείς, όσο και αν ακούγεται αυτό σκληρό, να μην περιορίσουμε το ενδιαφέρον μας στα εισοδήματα των εργαζομένων και να προσπαθήσουμε να δούμε την μεγαλύτερη εικόνα και μάλιστα οι μεγάλες ζημίες γίνονται από λίγα πλοία τα οποία έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Μας είπε ο κύριος Αρσένης ότι πάρα πολλά από τα λιεύματα τα οποία έτσι και αλλιώς ε, συλλέγονται δεν είναι βρόσιμα. Πάρα πολύ απλό. και εξέφρασε ανησυχίες ο κύριος Αρσένης και για τα κοραλιογενή και για τα σπογγοειδή και αυτά απαιτούν πάρα πολύ μεγάλους χρόνους, ε, τεράστιους χρόνους για να διασφαλίσουν την αναπαραγωγή τους και ταυτόχρονα δίνουν και τη δυνατότητα σε αλλιεύματα να κάνουν το ίδιο. Γνωρίζουμε φυσικά ότι τα παραγάδια δεν είναι πανάκια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα παραγάδια δεν είναι η καλύτερη λύση. Αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση η οποία να αφορά ακριβώς τους αλλιευτικούς εξοπλισμούς. Να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των αλλιευμάτων και σε βενθικές περιοχές. Και να προσπαθήσουμε επίσης ε, να βρούμε τρόπους να αλλιεύουμε τα είδη που μας ενδιαφέρουν να φάμε και όχι να αλλιεύουμε γενικά ό,τι κινείται. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Θα πρέπει να δούμε και για τα όρια του βάθους, τα οποία θα γίνονται αποδεκτά και για τα είδη των αλλιευμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καντέκ παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Κρήτονα για την δουλειά του. Δεν συμμερίζομαι, θα πω, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Θα προσπαθήσουμε μέσω των συναντήσεων και με τους κοιόδης εισηγητές να συνεννοηθούμε. Να θυμίσω όμως ορισμένα στοιχεία. Καταρχάς κάτι που υπόθηκε ήδη. Η πλειοψηφία των αλλιευμάτων των εμπορικών μια χαρά είναι. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτά. Είδαμε τι έγινε και με τα τάκ και τις ποσοστώσεις του 12. Σε ορισμένα είδη εμπορικά αυξάνονται τα τάκ. Ε, ταυτόχρονα τα στοιχεία τα επιστημονικά που έχουμε από το 12 δείχνει ότι η εκμετάλλευση των ε, αλλιευμάτων βαθέων ε, υδάτων έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο βιώσιμο σε σχέση με το τι είχε γίνει το 90. Το θέμα είναι περίπλοκο, δεν αμφιβάλλω. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στο λεγόμενο gel de l'empreinte, δηλαδή την ανείχνευση και τον καθορισμό του ίχνους. Να δούμε ε, ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες η κατάσταση έχει κλονιστεί λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και θα πρέπει επίσης να δούμε τι θα γίνει και με τη γενίκευση των ζωνών προστασίας των ευάλωτων περιοχών. Εγώ είπα στην αρχή ότι δεν συμφωνώ πλήρως με αυτά τα οποία είπε ο φίλος Κρήτον στα πλαίσια της εκθέσεώς του. Διαβάζοντας ε, την έκθεση του βλέπω ότι ξεπερνάει κατά πολύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να πω στη συγκεκριμένη φάση ότι το 23, η τροπολογία 23 είναι ιδιαίτερα ενδεικτική των προθέσεων του εισηγητή. Λέει ότι ε, μια τράτα η οποία πηγαίνει στα 400 μέτρα, τώρα στα 200 από ό,τι φαίνεται, είναι κάτι το οποίο θεωρείται ότι αλλιεύει σε πάρα πολύ ε, μεγάλα βάθη. Γιατί όχι τα 100 να είναι μεγάλα βάθη, τα 50 να είναι μεγάλα βάθη αν θέλετε. Δεν είναι αφαίρετο αυτό. Με ποιο τρόπο ε, ορίζουμε το βάθος ότι είναι ε, μεγάλο βάθος. Λοιπόν, αυτό ήταν λίγο αστείο, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο κείμενο, η συγκεκριμένη πρόταση δεν φύγει μόνο ε, ε, την αλληλεία σε μεγάλα βάθη, αλλά την αλληλεία με τράτες γενικότερα. Υπάρχει μια επιθυμία μεσοπρόθεσμης απαγόρευσης κάθε αλλιευτικής δραστηριότητας με τράτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις οικονομίες των παράκτιων περιοχών μας, γιατί τα περισσότερα από τα σκάφη μας σε μία στιγμή ή σε μία άλλη αλλιεύουν ακριβώς με τράτες, με μηχανισμούς τράτας. Θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν ότι τα παραγάδια θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ε, ε εν μέρη ε, τις τράτες. Όχι. Κοιτάξτε, στην περίπτωση αυτή που θα πληρώσουν το λογαριασμό στην περίπτωση αυτή είναι οι καρχαρίες σε υψηλά βάση αν χρησιμοποιήσουμε τα παραγάδια. Αν εμείς κυνηγάμε μια πεσκανδρίτσα και πιστεύετε ότι θα την πιάσουμε την πεσκανδρίτσα αυτή ή το βατραχόψαρο αν θέλετε με το παραγάδι πάρτε με τηλέφωνο εκτός, ε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση εκτός αν τροποποιήσετε το είδος εσείς της πεσκανδρίτσας ή του βατραχόψαρου. Το βατραχόψαρο ποτέ δεν θα τσιμπήσει ένα παραγάδι. Αν βρείτε εσείς κάποιον να το κάνει να μου το πείτε. Λοιπόν πέρα από αυτό, αυτό το οποίο έχει σημασία στην έκθεση η οποία παρουσιάζει ο κύριος Αρσένης είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τα παράπλευρα στοιχεία ηχθειοπληθυσμών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακριβώς είδη τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στα παραγάδια. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και σας έφερα το παράδειγμα των καρχαριών υψηλού βάθους, μεγάλου βάθους μάλλον και υπάρχουν και άλλα εδώ. Το θέμα είναι επίσης ότι επιβάλλουμε στα κοινοτικά σκάφη ε, συνθήκες αλληλείας που δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα μη κοινοτικά σκάφη. Θα απαγορεύσουμε δηλαδή να κάνουν πράγματα τα σκάφη μας που τα σκάφη της Νορβηγίας και της ε, Ισλανδίας θα κάνουν στις ίδιες περιοχές γιατί ξέρουμε ότι έχουν δικαίωμα να αλλιεύουν εκεί. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα λογικό. Ε, λυπάμαι που έφυγε η κυρία Ρόσβαχ. Κρίμα αλλά θα τις μεταφέρετε αυτά τα οποία είπα. Σέβομαι φυσικά τους συναδέλφους των υπολείπων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι συνάδελφοι όμως των υπολείπων επιτροπών δεν σέβονται πάντα τους συναδέλφους της δικής μας επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, λίγοι από αυτούς που είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται όταν συζητάμε. Ε, ε, ε, τα θέματα της αλίας. Δεν γνωρίζουν την προβληματική της αλίας. Και η ψηφοφορία που έγινε χθε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα μου επιτρέψετε όχι να την αμφισβητήσω γιατί δημοκρατικά ελήφθη η απόφαση. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι πήραν την απόφαση αυτή χωρίς να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, όπως και να έχουν τα πράγματα, θα ξεκινήσουμε σύντομα, προβλέπει τη Δευτέρα το απόγευμα, μια πρώτη συνάντηση δεν ξέρω αν την επιβεβαιώνει, ήδη θα συναντηθούμε δηλαδή μαζί με τον κύριο Αρσένη και θα προσπαθήσουμε, εφόσον μπορέσουμε βέβαια, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ευαίσθητο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκοζές, παρακαλώ. Euh, euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντίθετα με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, προηγούμενο ιδιαίτερα συναδέλφο, εγώ θα ενταχθώ αν θέλετε στη λογική του εισηγητή μας και θα ενταχθώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και όπως είπε ο κύριος Γκάλακερ, θα ήθελα να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν χώρο συνένεσης για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι επί της ουσίας Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχει σήμερα ο τομέας και η οικονομική δραστηριότητα που μας ενδιαφέρει, της αλίας δηλαδή, μια δύσκολη προσπάθεια έβρεσης ισορροπίας ανάμεσα στην πραγματικότητα, στη συγκυρία, την οικονομική και την κοινωνική και στις ανάγκες του μέλλοντος, οι οποίες είναι κυρίως οικολογικές και έχουν βέβαια συνέπειες οικονομικές και κοινωνικές. Καλούμεθα λοιπόν εμείς να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Τώρα, για την αλληλεία σε μεγάλα βάθη, θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Καταρχάς, να δούμε το παρόν, τη συγκυρία, τα οικονομικά συμφέροντα, τις θέσεις απασχόλησης που παρέχει ο τομέας και ταυτόχρονα να δούμε τις οικολογικές συνέπειες αυτής της οικολογικής δραστηριότητας, της οικονομικής συγγνώμη δραστηριότητας, σε επίπεδο οικολογικό, σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αν έχουμε καλή πίστη θα διαπιστώσουμε ότι γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ ισόρροπα ανάμεσα στο οικονομικό και στο οικολογικό κομμάτι. Απαιτείται λοιπόν να αλλάξουμε την κατάσταση, να βρούμε μια νέα ισορροπία και προς όφελος της ποιότητας των μεγάλων εν περιπτώσει περιοχών στις οποίες γίνεται η αλληλεία σε υψηλά βάθη, σε μεγάλα βάθη και προς όφελος της οικονομικής πραγματικότητας. Η αλληλεία αυτή είναι το 1% των αλλιευμάτων, 1% των αλλιευμάτων στον Ατλαντικό, στην περιοχή αυτή βέβαια. Τώρα, εγώ θα μιλήσω για τη γαλλική πραγματικότητα, γιατί δεν κατέχω την ισπανική ή την πορτογαλική πραγματικότητα, η οποία θα έλεγα ίσως είναι γειτονική. Ε, δέκα σκάφη γαλλικά ασχολούνται με αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Δέκα τράτες γαλλικές. Το 1% δηλαδή, το 1% κάτω από το 1% του γαλλικού αλλιευτικού στόλου. Και σε επίπεδο απασχόλησης, άντε να μιλήσουμε για 100 ναυτικούς και έμεσα ίσως άλλη τόση ε, στην επεξεργασία κτλ. Αν και θα πρέπει βέβαια να μην αγνοήσουμε και το κατανοώ αυτό, ότι αυτή η δραστηριότητα σε μεγάλα βάθη αφορά και κάποιους μικρούς αλληλείς, στους οποίους παρέχει μια συμπληρωματική δυνατότητα πρόσκλησης εισοδήματος. Τώρα, το οικονομικό κομμάτι λοιπόν, όπως σας είπα και όπως βλέπετε, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα όμως, δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τις θέσεις αυτής της απασχόλησης να τις αγνοήσουμε και να τις καταστρέψουμε κοιτώντα αλλού. Θα πρέπει στα πλαίσια των προτάσεων που θα κάνουμε να βρούμε λύσεις αλλαγής δραστηριότητας, λύσεις ε, πολλαπλών δραστηριοτήτων στο μέλλον για τις συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης. Αυτό για το παρόν, για το μέλλον τώρα, στο κομμάτι το οικολογικό. Έχουμε καταστροφικές συνέπειες της δραστηριότητας αυτής που αποδεικνύεται από το σύνολο των επιστημονικών συγχείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν θα τα επαναλάβω, τα είπε πολύ καλά ο κύριος Αρσένης. Είναι ιδιαίτερο ευάλωτοι οι ηχθειοπληθυσμοί. Είναι πάρα πολύ αργή η ανανέωση των, <coughs> των στόκ, των ηχθειοπληθυσμών πρέπει ε, να κλείνω λέει ο μιλητής και σε σχέση επίσης με την καταστροφή των οικοσυστημάτων τα οποία είναι αναντικατάστατα και σε επίπεδο ε, βιολογικό, βιοπικιλότητας κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία μας οδηγούν αναπόφευκτα συνάδελφοι να προσπαθήσουμε να μην πιέσουμε ιδιαίτερα αλλιευτικά τον τομέα ε, του μεγάλου βάθους. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το βάθος των ωκεανών δεν είναι το μέλλον της αλίας, γιατί η αλία η οποία ε, θα έλεγα εξελίσσεται σε αυτές τις ζώνες δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Ένα λεπτό μόνο και θα κλείσω. Ε, μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και μπροστά στις ευθύνες τις οποίες έχουμε, νομίζω ότι έχουμε πλέον την υποχρέωση να ξεπεράσουμε τα ημίμετρα, να ξεπεράσουμε τα συντηρητικά μέτρα όπως ε, το ε, πάγωμα ας πούμε, των ποσοτήτων κτλ. Νομίζω ότι όπως το συστήνει η Επιτροπή και όπως το συστήνει και ο εισηγητής μας να πάρουμε μια γενναία απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι σταδιακά να αποσύρουμε τις στράτες βάθους που α, είναι η πιο καταστροφική πρακτική σε σχέση με την ανανέωση ε, των συγκεκριμένων αλλιευμάτων. Τελειώνω εδώ ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε μια συγκεκριμένη τεχνική αλληλείας, όχι να απαγορεύσουμε την αλλιεύση συγκεκριμένων αλλιευμάτων. Το θέμα δεν είναι να σταθούμε παρανοϊκοί απέναντι σε μια πιθανή πλήρη απαγόρευση της τράτας. Όχι, κανένας δεν το θέλει αυτό. Πρέπει να στραφούμε όμως σε διαφορετικές εναλλακτικές δραστηριότητες όπως και η μετατροπή της τράτας σε παραγάδι. Σας ευχαριστούμε κυρία Φράγκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό το θέμα όπως των καρχαριών είναι πολύ έντονα με απήχηση στον τύπο θέματα και θα ήθελα να είμαστε σε θέση εμείς εδώ στην Επιτροπή Αλίας να καταλήξουμε σε συνετές θέσεις, λογικές θέσεις, εκτός πίεσης ε, και έντασης που υφιστάμεθα όλοι πολλές φορές και μάλιστα έντονης πίεσης. Αυτό πρώτο. Δεύτερο. Και αυτό το οποίο είπε η κυρία Ρόσμπαχ. Φαίνεται όπως ότι εδώ σε αυτό το θέμα όλα αλλιεύονται παντού χωρίς καμιά ρύθμιση και πρέπει σίγουρα να δούμε ότι αυτό δεν είναι από τα αλήθες. Η βαθιά η στα βαθιά νερά ρυθμίζεται από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Έχουμε όλη, όλο το σύστημα προστασίας των ευαίσθητων ε, ε, βιοτόπων. Δεν θέλω να πω ότι έγιναν όλα, αλλά έχουν γίνει πράγματα. Στην ακρόαση που κάναμε εδώ, ιδιαίτερα οι επιστήμονες που είχαν έρθει, μας είπαν με κάθε σαφήνεια ότι αυτή την τελευταία δεκαετία μετά τα όσα είχαν γίνει και ήταν οι ε, υπερβολές ε, κατά την προηγούμενη δεκαετία υπήρξε μείωση 50%. Επαναλαμβάνω, μείωση 50% της αλληλευτικής προσπάθειας. Και ποια ήταν η απόρρια αυτού του μέτρου. Η απόρρια θα ήταν ότι τα κύρια τρία κυριότερα αλλιεύματα που είναι ε, το, το βατραχόψαρο και το Ντρόψαρο θα ε, βρισκόντουσαν στην ε, ίδια κατάσταση που είχε ανακάμψει. Αυτό μας είπαν εδώ οι επιστήμονες που είχαν συμμετάσχει στην ακρόαση. Δεν είπα τίποτα άλλο. Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα ίδια να πω ότι δεν είναι όλα τα είδη σε μια τέτοια αρνητική κατάσταση. Υπάρχει ανάκαμψη αλλιευμάτων. Φυσικά όταν λέτε εσείς ε, κύριε Ασένη από την άλλη πλευρά ότι τα είδη βαθ βαθιάς, ε, βαθαίων υδάτων ε, ε, είναι με αυτόν τον τρόπο απειλούμενα. Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και επίσης αναφέρθηκε εδώ ότι για αυτό το ψάρι το οποίο έχει μικρότερη περίοδο βίου από 30 χρόνια. Γι' αυτό μας είπε ο κύριος Φίσερ ότι ήταν διαφορετική κατάσταση. Για τα 30 χρόνια και η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ήταν θετική για αυτά τα είδη. Γι' αυτό λοιπόν να μην συγχαίουμε εδώ όλα αυτά τα πράγματα σε σχέση με τους ε, καρχαρίες ε, λέγοντας ότι όλα τα είδη καρχαριών βρίσκονται στο ίδιο, στην ίδια κατάσταση και να συγχαίουμε τα πράγματα. Τα τρία κυριότερα αλλιεύματα αυτών των βαθαίων υδάτων βρίσκονται σε ανάκαμψη, σαφώς, και βρίσκονται ακριβώς σε αυτό το όριο το οποίο έχει επιτευχθεί. Αυτό μας το είπαν επιστήμονες με τεκμήρια εδώ στην Ακρόαση. Να μην λέμε πράγματα λοιπόν τα οποία δεν ευσταθούν, δεν αληθεύουν. Το θέμα των 200 μέτρων ως όριο τώρα, το περιβόητο αυτό θέμα, ε, ο εκπρόσωπος μας είπε σαφώς ότι στον ορισμό αυτό ακριβώς ήταν εφικτό έπρεπε να καθοριστούν ήδη βαθαίων υδάτων που κατά 50% της βιομάζας τους βρίσκονται κάτω από ε, τα 200 μέτρα. Όλα αυτά βέβαια ε, συγκρούνται με άλλες ε, διατάξεις που έχουμε. Μετά από αυτό θα ήθελα να πω κάτι για την ε, κοινωνική, κοινωνική οικονομική συμφωνία και σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Αρσένης. Δεν αληθεύει ότι αυτό αφορά λίγα σκάφη. Δεν αληθεύει. Διότι εδώ αναφέρονται κάποια από τα στοιχεία τα οποία στοχεύουν σε σκάφη που έχουν μόνο αποκλειστικό στόχο τα είδη βαθιάς θάλασσας. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι θα δεχθούμε και εκείνα τα σκάφη που παρεμπίπτοντα αλλιεύματα έχουν μόνο από τα βαθιά νερά. Το θέμα είναι πολύ ευρύτερο λοιπόν, πολύ ευρύτερο και σε σχέση με τις επικρίσεις που σε σχέση με την μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν λαμβάνεται λέει υπόψη η οικονομική κοινωνική πραγματικότητα και το εύρος και οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε. Χωρίς να το ε, είμαι εγώ η οποία τα λέει όλα αυτά, διότι μπορεί να είναι ριζοσπαστικές κάποιες ε, δικές μου ε, η προηγούμενη έκθεση που έκανε η Γενική ε, ε, το Τμήμα Μελετών ε, επισημαίνει ότι μία από τις κύριες επικρίσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι δεν ελήφθη υπόψη η κοινωνική, οικονομική επίπτωση αυτών των μέτρων. Και θα το πω και στα αγγλικά για να μην το κάνω λάθος. Δηλαδή η ε, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μελετά ακριβώς αυτά τα θέματα έκανε αυτές τις ε, ε, διατυπώσεις με επικρίσεις ήδη χρόνια πριν για ένα τέτοιο λοιπόν σημαντικό θέμα πώς μπορεί να αναφέρεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν αληθεύουν τα στοιχεία σε σχέση με την Ισπανία. Δεν λαμβάνουν υπόψη εκείνα τα σκάφη που έχουν παρεμπίπτοντα αλλιεύματα από τα βαθιά ύδατα. Είναι λοιπόν παραλογισμός ε, να, να λέγεται ότι δεν ελήφθη υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εύρος του προβλήματος. Το λέω εδώ ανοιχτά και ξεκάθαρα και σε σχέση με τις ΜΚΟ. Αυτό πρέπει να ακουστεί ως παρατήρηση. Και τώρα το θέμα των ε, ε, παραγαδιάρικων ή το θέμα των ε, τρατών βυθού. Πρέπει να πούμε ότι οι επιστημονικές μελέτες πρέπει να δούμε τι λένε. Το Ίδρυμα Οκεανογραφικών Μελετών συνέταξε μια μελέτη που δείχνει ότι πάνω από 80% των συνολικών αλλιευμάτων είναι καρχαρίες βαθέων υδάτων. Λοιπόν δεν είναι τόσο απλά τα θέματα όπως παρουσιάζονται και υπάρχουν και πολλά είδη τα οποία δεν είναι δυνατόν να να αλλιευθούν ε, με αυτόν τον τρόπο, ε, λέγει η κυρία Φράγκα, όπως ε, ανέφερε ο εισηγητής. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν με το ένα είδος και το άλλο. Δεν λέω ότι η γρήπη, οι τράτες και τα παραγαδιάρικα είναι το ίδιο. Ξέρω ότι η γρήπη, τα παρα... οι τράτες μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Ωστόσο, σε λασπόνερα δεν μπορεί να κάνει καμιά ζημιά ο γρήπος. Πρέπει να δούμε αυτό και να το διαφοροποιήσουμε. Όχι, δεν ολοκληρώσα, Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω ολοκληρώσω ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ωραία, ολοκληρώστε. Μια ολόκληρη σειρά μέτρων λοιπόν έχουμε εδώ. Τι γίνεται με την επικέντρωση σε σχέση με τα ευάλωτα, ε, με τους ευάλωτους βιοτόπους ε, της θάλασσας. Θα μπορούσαμε να επιλύσουμε απόλυτα το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αν λαμβάναμε αυτό υπόψη. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας αφαιρέσω τον λόγο, αλλά έχουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και πρέπει να μπορέσουμε να ε, συγκεράσουμε τα πράγματα γιατί διαφορετικά δεν θα φτάσει ο χρόνος. Ο χρόνος πιέζει. Ο κύριος Μιλάνα παρακαλώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, τηλεγραφικό. Πρώτο τηλεγράφημα. Ο Κρήτον έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια με ένα υψηλό αίσθημα ευθύνη. Δεύτερο τηλεγράφημα. Νομίζω ότι η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι λανθασμένη. Συζητάμε για τα συμπεράσματα της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και όχι τις προτάσεις του Κρήτονα. Τρίτο τηλεγράφημα. Τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα που θέτει ο Κρήτον. Εκπλήσωμαι γιατί κάποιοι από τους συναδέλφους θεωρούν σημαντικό σήμερα να υπερασπιστούν ακριβώς τους καρχαρίες ε, μεγάλου βάθους. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Μακάρι να γινόταν αυτό κάθε φορά που συζητάμε τα της αλίας. Τέταρτο. Εκπλήσωμαι ότι ανησυχούμε επίσης για το στόλο μας, και το έλεγε ο Αλά εδώ, το οποίο έχει προβλήματα ανταγωνιστικότητας με άλλες χώρες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Το λέω αυτό εδώ και τέσσερα χρόνια για τον κανονισμό για τη Μεσόγειο όπου οι ίδιοι οι κανόνες γίνονται σεβαστοί από 8 μεσογειακές χώρες και δεν γίνονται σεβαστές από 14 ε, μεσογειακές χώρες. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχετε συστηματικά όλοι αγνοήσει παρόλα αυτά. Τελευταία παρατήρηση. Είμαι αισιόδοξο. Εγώ νομίζω ότι η αντικειμενικότητα με την οποία έθεσε το θέμα και ο Σαρσένης και ο διάλογος τον οποίο έχει ξεκινήσει, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω το σύνολο των πολιτικών μας θέσεων, θα μας οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Και τελευταίο πάλι, λέει για τρίτη φορά ο Μιλτής, ανησυχώ από το ότι ε, θα καθυστερήσουμε από ό,τι φαίνεται και ότι έχουμε να κάνουμε θα έλεγα με μια θα έλεγα υποβόσκουσα προσπάθεια να οδηγηθούμε στο θέμα ακριβώς ε, το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι στο θέμα το οποίο έχουμε εμεί θέσει εδώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκαν τα τηλεγραφήματα. κυρία Τόμας παρακαλώ. Oui, merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κρήτονα για την προσπάθειά του. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι έχει ξεκινήσει από ένα κείμενο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό. Το κείμενο της Επιτροπής δεν μας βοηθά. Έχουμε μια δύσκολη εξίσωση μπροστά μας σε σχέση με μια αλλιευτική δραστηριότητα. Θα έλεγα έχουμε τρεις αγνώστους εδώ. Πρώτον θέλουμε πράγματι να διασώσουμε το αλίευμα. Δεύτερον θέλουμε να διασώσουμε τα ευάλωτα οικοσυστήματα και τρίτον να προστατεύσουμε την οικονομία των παρακτήων περιοχών και τις θέσεις απασχόλησης. Να πω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει, και το λέω στον Ζαν Κλόντ, ε, το 1% των αλλιευμάτων ή ένα μικρό αριθμό, εν πάση περιπτώσει, σκαφών. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε την μελέτη κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων που απαιτείται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι αριθμοί που έχουμε είναι διαφορετικοί από αυτούς που είπε ο Ζων Κλοντ. Πράγματι, στη Γαλλία έχουμε 100 ναυτικούς. Ένας ναύτης όμως, ένας ναυτικός σημαίνει άλλες 6 θέσεις απασχόλησης ε, στην ε, ξηρά, στην υπηρετική χώρα. Οπότε μιλάμε για 600 και ιδιαίτερα στην πόλη του Λοριόν έχουμε 600 θέσεις απασχόλησης που ε, απασχολούνται ακριβώς και αυτή είναι, ε, αυτό είναι στοιχείο που δίνει ο Δήμος του Λοριό. Και δεν, ε, δεν ασχολούμεθα καθόλου και δεν γνωρίζουμε το μέγεθος των υπολείπων βιοτεχνικών μορφών αλληλείας που συμπληρωματικά ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα. Είπαμε λοιπόν στόχος η προστασία του είδους, στόχος η προστασία του περιβάλλοντος, στόχος η προστασία των θέσεων απασχόλησης. Το εύκολο θα ήταν να προκρίνουμε το ένα εις βάρος των άλλων. Σε αυτή την περίπτωση ε, θα μπορούσαμε να τα απαγορεύσουμε όλα, τα πάντα όλα όπως λέμε. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε στον κόπο να βρούμε μία λύση και γι' αυτό παίρνουμε όλα τα προστατευτικά μέτρα και δεν κάνουμε τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να εκπλησόμεθα αν η Ευρώπη περάσει στην ύφεση. Αυτό το οποίο εγώ προτείνω είναι ένας προσανατολισμός ο οποίος προσπαθεί να λάβει υπόψη και να συνδυάσει τα τρία αυτά στοιχεία, προστασία του είδους, προστασία των ναυτικών οικοσυστημάτων, των θαλασσίων συγγνώμη, οικοσυστημάτων, που δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται παντού με τον ίδιο τρόπο και προστασία των θέσεων απασχόλησης. Έχει δίκιο ο Πάτρε Κόουπ που είπε ότι ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να απαγορεύσουν και σε αυτούς που θέλουν να βρουν μια ισορροπημένη λύση θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη δεύτερη πρόταση. Μετά από την ακρόαση που κάναμε με τους εμπειρογνώμονες και τους επιστήμονες, βρήκαμε στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και στη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τελικά δεν ε, ελήφθη υπόψη. Καταρχάς το λεγόμενο πάγωμα του ίχνους, σε σχέση με την επιφάνεια των, του, <clears throat> η επιφάνεια του βυθού. Δεν θα πρέπει να θέσουμε τώρα συνολικά την προβληματική ε, της στράτας. Νομίζω όμως ότι σε σχέση ε, με τις πιθανές δυσκολίες που υπάρχουν για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι μπορούν να ξεπεραστούν. Και ε, νομίζω ότι δεν πηγαίνουν σε άλλου είδους ε, εδάφη βυθού θα έλεγα οι τράτες παρά μόνο σε αυτές που δεν τους προκαλούν βλάβες. Δεν θα πάνε σε βραχώδεις βυθούς σαν παράδειγμα. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που μίλησαν για αυτά τα οποία είπε ε, η συνάδελφος από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και της το είπα την ώρα που έφευγε. Θα έπρεπε να πάρει μέρος σε αυτή τη συζήτηση, γιατί η ψηφοφορία της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχει μεγάλο βάρος. Αντίθετα με αυτά που είπε, το πρόβλημα δεν είναι τα αλλιεύματα, γιατί είναι σταθεροποιημένα τα αλλιεύματα. Αν και μπορούμε να βελτιώσουμε βέβαια την, πίεση που ασκείται στα αλλιεύματα. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ και απευθύνομαι στον Κρήτονα. Ας, ας σταματήσετε να επιμένετε με το, φόβητρο των 200 μέτρων. Κοιτάξτε, τα 200 μέτρα κρύβουν άλλα προβλήματα. Το θέμα το οποίο τίθεται στη συγκεκριμένη περίπτωση έμεσα είναι η απαγόρευση της τράτας και ας μη σαλαποποιούμε τα πράγματα. Σήμερα δηλαδή ας κόψουμε την τράτα ε, σε μεγάλο βάθος, αύριο ας κόψουμε την τράτα σε μεσαία βάθη και μεθαύριο ας κόψουμε και τα παραγάδια ακόμα. Δεν πάει έτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα όπως πρέπει και είναι θέμα καλής συμπεριφοράς κοινοβουλευτικά Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αρσένη που εκπώνησε αυτή την έκθεση από πλευράς του. Τώρα δεν ξέρω να πω αν ε, με αυστηρότητα ή όχι, διότι υπήρχε πολύ μικρός χρόνος γι' αυτό και το γνωρίζει και ήταν, είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο πρέπει διαρκώς να επαναλαμβάνουμε αυτό αυτή την κατάσταση στο σώμα. Αληθεύει όμως ότι οι όροι υπό τους οποίους εργαζόμαστε οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές με τον πολύ περιορισμένο ελάχιστο χρόνο που έχουμε δεν φτάνουν έγκαιρα τα έγγραφα δεν θέλω να πω ποιο είναι ο τελικά υπεύθυνο ε, για το αν φτάνουν ή όχι έγκαιρα οι εκθέσει στα χέρια μα. Το ζήτημα όμω είναι ότι γι' αυτό το έγγραφο, αυτό το είχαμε στα χέρια μα μόνο μια εβδομάδα στα αγγλικά και δύο μέρε όλε και όλε στα ισπανικά. Έχουμε όμως μήνες που αντέχουμε την πίεση του ενός ή του άλλου που μας λένε τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε. Και θα πρέπει να πούμε σε ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κοινοβούλιο τέτοιου είδους καταστάσεις και πιέσεις δεν ωφελούν κανένα. Ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Πρέπει να έχουμε κοινή ευθύνη όλοι και ισοδίκαια να αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Και πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια ρυθμιζόμενη αλία. Πρόκειται για ένα κανονισμό που πραγματικά θα έπρεπε, μια και είναι πολύ πρόσφατος, να είχε γίνει μια μια αξιολόγηση Προτού υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να είχαμε μια τέτοια αξιολόγηση προτού έχουμε μια νέα πρόταση σαν αυτήν εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη ριζοσπαστικότητα, ε, συγχωρέστε μου την ε, έκφραση, θα έπρεπε να έχουν γίνει τα πράγματα σωστά πιο πριν, όπως θα έπρεπε, δηλαδή με σύνταξη μελέτης επιπτώσεων. Είμαι υπερήφανη για το ότι η χώρα μου είναι η μόνη που το 2005 για να προστατευτούν τα ευάλωτα οικοσυστήματα και επίσης είναι αυτονόητο τα είδη που ζουν σε βαθιά ε, νερά και απειλούνται με εξαφάνιση, ξεκίνησε η χώρα μου με επαΐοντες επιστήμονες ε, με ένα εγχείρημα που έδωσε σημασία στην εντολή των Ηνωμένων Εθνών που είχε ως αίτιο την διατύπωση και ανείχνευση νέων περιοχών κινδύνου από τους επιστήμονες και για τα είδη. Και αμέσως υπήρξαν μέτρα τεχνικά που ελήφθησαν και σχέδια ανάκαμψης για τα αλλιεύματα. Παρόλα αυτά τα οποία έγιναν από πλευράς μας δεν είναι αυτό το οποίο δείχνει ποια είναι η πραγματική κατάσταση των πραγμάτων, αλλά δείχνει πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα σε σχέση με την βιοπικιλότητα που θέλουμε να διασφαλίσουμε στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε ε, αιφόρα αλλιεύματα, αηφόρο αλλιεία που να μπορεί να διατηρηθεί και πρέπει να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία, αυτές οι εκθέσεις οι επιστημονικές που αν μπορεί κανείς να τις δει και από πλευράς ε, των ε, επιστημονικών συμβουλευτικών οργάνων τον ε, ΡΑΚ όσον αφορά τα νοτιοδυτικά ε, ύδατα για παράδειγμα έχουμε απόψεις που διατυπώνονται και δεν υπάρχουν κάποιες, δεν υπάρχουν κάποιες κοινέ προτάσεις ή συστάσεις γιατί δεν υπάρχει μια κοινή θέση. Τι θέλω να πω. Είναι ένα θέμα επαρκώς σημαντικό και θα έπρεπε με την επαρκή σοβαρότητα να το είχαμε αντιμετωπίσει, να το αντιμετωπίζαμε ώστε σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος που ψήφισε δεν υπήρξε καμία ε, πρόσκληση ε, έχουμε πάντα και ε, επικοινωνία και ε, μηνύματα σε σχέση με τις συναντήσεις και συνεδριάσεις. Ούτε ζητήθηκε σε σχέση, για παράδειγμα, να υπάρξει κάποια γνωμοδότηση ή τοποθέτηση από πλευρά μας. Ας είμαστε αυστηροί και δίκαιοι. Αυτό που είχαμε είναι πολύ λίγος χρόνος και παραπονούνται οι επιστήμονες ότι δεν υπήρξε χρόνος για να συντάξουν μια έκθεση. Δεν μπόρεσε να υπάρξει μελέτη επιπτώσεων. Δεν υπήρξε τέτοια μελέτη. Λοιπόν, δεν έχουμε εδώ μία, ας το μία θέση υπεράσπισης ε, ε, σε σχέση που ε, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος που εγώ θέλω να προστατέψουμε την κοινοβουλευτική μου ομάδα καταλήξαμε στο να διαρωτόμαστε αν είμαστε συνεκτικοί στο τέλος τέλος με τις θέσεις μας ή όχι. Πιστεύω ότι εδώ ο Αρσένης που έκανε την δουλειά όπως έπρεπε θα έπρεπε να το μελετήσουμε νυφάλια να υπάρχει περίοδος αξιολόγηση για την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Είναι πολύ σύντομη, πολύ πιεστική η προθεσμία αυτή. Με του περιορισμού που εργαζόμαστε εδώ, όλο με πιέσει ε, που αντιμετωπίζουμε εργαζόμαστε υπό τεράστια πίεση και με πολύ στενές ε, χρονικές περιόδους ως προθεσμίες ή διορίε. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος θα ζητούσα να ληφθούν όλα αυτά υπόψη και αν είναι δυνατόν κάτι να γίνει να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, να έχουμε μεγαλύτερο χρόνο εργασίας ως Εύρος για να μπορέσουμε πιο άνετα, ε, σε μεγαλύτερο βάθος να δουλέψουμε. Θέλω να αναφέρω και να υπογραμμίσω την ε, θέση μου. Είμαι υπέρ πάντα αυτών που υπερασπίζαμε, ότι οι τελευταίοι έχουν λιγότερο χρόνο στην παρέμβασή τους δυστυχώς. Είμαστε σε σχέση με την προστασία απόλυτης προστασίας, υπέρ απόλυτης προστασίας με τους βιοτόπους και την συνεκτικότητα αυτών των προσπαθειών προστασίας του περιβάλλοντος ε, όσον αφορά τα ευάλωτα είδη. Υπάρχουν τεχνικά μέσα και ε, δυνατότητες που άρχισαν να λειτουργούν στη χώρα μου, που άρχισαν να είναι υποφελή. Πρέπει να τα μελετήσουμε όλα αυτά, όλα. Να τα μελετήσουμε και να μπορέσουμε να δούμε ε, τι μπορεί να γίνει. Να εξετάσουμε το πράγμα από όλε τι πτυχέ δεν είναι το θέμα να είναι κανείς πιο πράσινος, ε, πιο ε, γαλάζιος ε, ή πιο πορτοκαλής. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ρέντις παρακαλώ. Yes, Davis. Uh, Davis, Ντέιβις. Davis. Davis παρακαλώ, όχι Jenkins. Um, Πρόεδρε. Συμβαίνουν ε, ταυτόχρονα διάφορα συνεδριάσεις επιτροπών, πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε διαφορετικές ε, ατζέντε, διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Πιστεύω ότι όλοι εδώ στην Επιτροπή Αλίες θέλει να σταματήσει η μη αηφόρος αλία και οι μη αηφόρες πρακτικές της αλίας που ζημιώνουν το θαλάσσιο περιβάλλον ή τα αλλιεύματα ε, και επιφέρουν ζημίες οι οποίες είναι αδιόρθωτες, δεν μπορούν ποτέ να ε, διορθωθούν και να επανέλθουν τα αποθέματα. Η δική μου ισορροπία την οποία επιδιώκω είναι η εξή. Δεν θέλω να δυσκολέψω τη ζωή περαιτέρω των ε, αλλιέων που ψαρεύουν στα νερά αυτά, αλλά των οποίων ο στόχος δεν είναι τα ψάρια των βαθέων υδάτων. Και όμως ε, αθέλητα πιάνουν τέτοια ψάρια. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις και πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μια ισορροπία στις προτάσεις, ώστε αυτοί οι κατά λάθο αλληλείς βαθέων υδάτων δεν φύγονται, δεν ζημιώνονται. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εχθές Ξέρετε ότι η Επιτροπή υπερψήφισε ε, την ε, πρόταση της Κομισιόν και της κυρία Ράουσενμπεργκ με 58 εναντί μια ψήφου κατά. Ε, τώρα, Πρόεδρε, το κοινό, οι πολίτες μας στην Ευρώπη πιστεύουν ακράδαντα ότι δεν έχουμε ιδέα τι κάνουμε εμείς. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι πολύ δύσκολο να τους πείσουμε ότι υπάρχουν όντως μέλη του Κοινοβουλίου που γνωρίζουν την κατάσταση και που θέλουν να ψηφίσουν μέτρα για την προστασία των αλλιέων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε το σωστό. Στην Επιτροπή μου εχθές η μεγαλύτερη μου ανησυχία ήταν αυτό το βάθος, το όριο του βάθους. Η Κομισιόν πρότεινε ότι ορίζεται το βάθος αυτό από τα αλλιεύματα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος προτείνει ένα αριθμητικό όριο βυθού ορισμού της αλίας βασέων υδάτων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό, να πάρουμε δηλαδή ένα μέτρο και να αρχίσουμε να μετρούμε το βάθος του ωκεανού. Δεν θέλω όμως να πιάνονται κατά λάθο στα δίκτυα και τα ψάρια αυτά που συνήθως βρίσκονται ε, στα βασιά νερά. Εχθές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν το δέχτηκαν, δεν δέχτηκαν αυτή την προσέγγιση και η Φιλελεύθερη ήταν η μόνη πολιτική ομάδα που είχε αντιρρήσει σε αυτό το μετρήσιμο βάθος της βασιάς αλίας. Εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν και πρέπει να βασιστούμε στο είδος των ψαριών στο... και όχι στο βάθος. Σας ευχαριστούμε. Σάντσες Περθέντο, πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής. Να πω ότι συμμερίζομαι το στόχο να προστατεύσουμε τα ευάλωτα είδη και τη βιοποικιλότητα που πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τα επαρκή μέτρα για αυτή την λειτουργία. Όχι να χρησιμοποιήσουμε πριόνι, αλλά να είμαστε προσεκτικοί με τα μέτρα που θα λάβουμε και αναλογικοί στη χρήση μας. Και για τα είδη πρέπει να δούμε ποιες επιπτώσεις έχουν στις κανονικές αλλιευτικές δραστηριότητες και ποιε επιπτώσει υπάρχουν σε αυτά τα ίδια οι αλληλευτικέ δραστηριότητε. Πολλέ φορέ δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει και πρέπει να έχουμε, να συναγάγουμε σωστά τα συμπεράσματα για τι αλληλευτικέ δραστηριότητε. Πρέπει κάποια πράγματα να διευκρινιστούν. Σε αφορά τι ζώνε, πιστεύω το ίδιο ισχύει όπω και στην ε, ε ξηρά. Υπάρχει ε, το θέμα τη ε, βιοπικιλότητα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να, είμαστε, να διαφοροποιήσουμε τα πράγματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Να ξέρουμε και τι κοινωνικο-οικονομικέ επιπτώσει που θα έχουν τα μέτρα ώστε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Αυτές οι πτυχέ πρέπει να ληφθούν υπόψη και από τους και από του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πρόεδρο. Η Επιτροπή λαμβάνει τώρα τον λόγο παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα σύντομα να απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις που τέσκαν και να να τη σχολιάσω κιόλα, σχολιάσω ορισμένα στοιχεία που δόθηκαν. Πόσα ε, αλλιευτικά σκάφη θα θίγονται από αυτές τις προτάσεις και ποιο είναι, ποιες είναι οι επιπτώσεις. Επαναλαμβάνω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι να ορίσει την αλληλεία βασέων υδάτων με μία σειρά από έναν κατάλογο ειδών, ψαριών, δεν έχουμε κανένα μετρήσιμο βάθος ε, ως βάση της προτάσεως μας, ούτε 200 ούτε 400 μέτρα. Εμείς ε, στοχεύουμε ε, ένα συγκεκριμένο αριθμό ειδών, αλλιευμάτων. Τώρα έχουμε λάβει υπόψη όλα, όλες, όλα τα αλλιεύματα, είτε είναι τα κύρια αλλιεύματα, είτε τα παράπλευρα τα παράπλευρα. Έχουμε λοιπόν υπολογίσει τα ποσοστά των ε, αλλιευόμενων ψαριών στο Βόρειο Ατλαντικό και έχουμε υπολογίσει το, τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε μετρήσει. Αλλιεύματα, εκφορτώσεις, οικονομικό κόστος, οικονομικά στοιχεία. Βεβαίως, είναι σωστό ότι ορισμένες αλλιευτικές κοινότητες στήγονται περισσότερο από άλλες και ξέρουμε ποιες είναι. Ε, σε ορισμένα παράκτια μέρη στην Γαλλία, στις Αζόρες, στη Μαδέρα και ε, βεβαίω χρειάζονται μέτρα, ορισμένα μέτρα. Αλλά ε, οι επιπτώσεις είναι αυτές που ήδη έχω εκφράσει και τις ξέρετε. Παρεπιπτόντος, το Κοινοβούλιο της Μαδέρας έχει εκφράσει την υποστήριξη της πρότασής μας, διότι πιστεύει ότι έτσι προστατεύονται τα αλλιευτικά τους αποθέματα. Η συζήτηση εδώ δεν ε, βασίζεται στις τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά βεβαίως σωστό. Εάν τεθεί ένα όριο 200 μέτρων, θα αλλιεύονται πολύ περισσότερες, πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ψαριών. Αλλά και πάλι, εδώ αποκλίνουμε από την πρόταση της Κομισιόν. Εμείς, η Κομισιόν, έχουμε προτείνει συγκεκριμένα αλλιεύματα, συγκεκριμένα είδη. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και ειδική αλληλεία και μία αλία. Παραδείγματο χάρη μπορούμε να πιάσουμε πεσκανδρίτσα, μπορούμε να πιάσουμε άλλα ψάρια ε, σε βαθιά νερά και μπορούμε να αποφύγουμε συγκεκριμένα είδη τα οποία δεν θέλουμε να πιαστούν. Ε, επίσης υπάρχουν μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στα διεθνή ύδατα. Το ISIS έχει κάνει μία αξιολόγηση των ε, μέτρων που εφαρμόζονται στη Βασιά Αλία, ιδιαίτερα το, τα μέτρα που ονομάζονται στα αγγλικά move on rule, δηλαδή πήγαινε παρακάτω, ο κανόνας του φύγε από εδώ και πήγαινε παραπέρα. Και αυτό ο κανονισμός λέει ότι αν χτυπήσει ε, ένα κοραλιογενή σπονγκοειδή ύφαλο, πρέπει να σηκώσει τα δίκτυα σου και να πας παραπέρα, να μετακινηθεί το σκάφος ένα-δύο μίλια, ναυτικά μίλια. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα συμπεράσματα του ISIS ε, του 2012, ε, μία από τις προτάσεις και προτείνει και τεχνικά μέτρα όπως προτείνουμε και εμείς για να αμβλυνθούν οι ανητικές επιπτώσεις. Υπάρχουν πραγματικά μεγάλο ποσοστό αλή, βασιάς αλίας που γίνεται στις, στα διεθνή ύδατα. Και γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Και να σχολιάσω αυτά που ελέγχθησαν. Καταρχάς το, το καθεστώς των αποθεμάτων. Το ISIS έχει συστήσει ότι ορισμένα αποθέματα, ληφτικά αποθέματα μπορούν να λιευθούν. Μπορεί να γίνει εκμετάλλευση σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, ως ενός ορισμένου βαθμού. Αυτό θα ωφελήσει τους αλείς που αλλιεύουν αυτά τα είδη. Αλλά ο πρόεδρος του ISIS σε μία ημερίδα εργασίας έχει πει σε, εδώ μέσα στην Επιτροπή αυτή ότι τα, τα αλλιεύματα είναι 20-30% αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν παλαιότερα, αλλά επισημεί να φτάσουν στο 50% ώσπου να δώσει το πράσινο σήμα για την επιτρεπόμενη εκμετάλλευση. Είναι λοιπόν εδώ και πάλι ένα, ένας μικρός αριθμός ε, αποθεμάτων, δεν καλύπτουν τα μεγάλα εμπορικά αλλιεύματα, αλλά ένα πολύ μικρό ε, αριθμό ε, αλλιευμάτων στα βασιά ύδατα. Και ένα άλλο σχόλιο που ακούστηκε αρκετές φορές, ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το ίχνος, διότι Παραδείγματο χάρη πολλοί λένε ότι στο λασπόδι βυθό δεν μπορούμε να καθορίσουμε το, τα ίχνη, το ίχνος. Ε, αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό εάν, χρησιμοποιήσετε τα δικά μας μέσα, τα δικά μας εργαλεία, μπορείτε και εκεί και σε αυτές τις περιοχές του βυθού να βρείτε τα είδη και αν ε, κάνετε ένα μοντέλο ε, για τα ευάλωτα είδη και τα οικοσυστήματα και τα είδη που πρέπει να προστατευθούν, θα δείτε επίσης ότι αυτό αφορά και περιφέρειες ε, του... Listen to the βραχόψαρου. Το αποτύπωμα λοιπόν μπορεί να βρεθεί, μπορεί να βρεθεί και μπορεί να μετρηθεί. Και τέλος ελέγχθη ότι η Κομισιόν δεν διαβουλεύτηκε, δεν έκανε την πρέπουσα διαβούλευση. Η STCF ε, ε, είναι η δική της επιστημονική επιτροπή σας πενθυμίζω λοιπόν ότι από το 2009 ζητήσαμε από την STCF που είναι η επιστημονική τεχνική ομάδα, συμβουλευτική ομάδα να μας παρουσιάσει ε, εξέσεις ε, ε, για τα θέματα αυτά. Όλες αυτές οι συστάσεις της STCF είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και έχουμε επίσης διαβουλευθεί εκτενώς με τα RAGS, τα περιφερειακά συμβουλευτικά κοινοβουλευτικά συμβούλια, τα, τα περιφερειακά συμβούλια και Επίσης έχουμε κάνει συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τα εκτελεστικά όργανα αυτών των φορέων. Άρα λοιπόν διαβουλεύσεις έχουμε κάνει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε κύριο Σαρσένης για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κάποιες απαντήσεις από την πλευρά μου σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν. Ε, τέθηκε από κάποιους συναδέλφους αν υπάρχουν ήδη επαρκή υφιστάμενα μέτρα. Όσον αφορά τα vulnerable marine ecosystems, τα ευαίσθητα ε, θαλάσσια οικοσυστήματα, θέλω να επισημάνω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα απολύτως μέτρο για την προστασία των σουγκαριών στον νοτιοανατολικό Ατλαντικό. Επίσης επανελήφθηκε ή υπόθηκε την Επιτροπή αλλά νομίζω ότι αξίζει να επαναληφθεί. Ε, στα, στις αιτιάσεις των συναδέλφων από το EPP, του κύριο Καντέκη και της κυρίας Φράγκα, ότι στην ουσία πάμε καλά. Τα ηχθοποθέματα ε, στην, ε, στε, βαθιά ε, είναι στην, ε, βελτιώνεται η καταστασή τους, έχουμε την επαναφορά τους σε βιώσιμα επίπεδα. Αυτό που έγινε και ήταν η εισήγηση του ISIS για πρώτη ε, φορά μόνο αυτά τα δύο τελευταία χρόνια για τα τρία αυτά είδη που αναφέρθηκαν είναι ότι το ISIS είπε ότι αυτά τα είδη σταθεροποιούνται σταθεροποιούνται απλά στα επίπεδα 20 με 30% της αρχικής βιομάζας. Σταθεροποιούνται δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο της βιομάζας τους. Τώρα, ε, ο κύριος Κατέκα αναφέρθηκε στο Monkfish. Ε, προφανώς το Monkfish δεν είναι ε, είδος βαθιάς θάλασσας, δίψης πίσης. Και είπαμε ότι οτιδήποτε αφορά είδη τα οποία επηρεάζονται ε, από αυτές τις προτάσεις. Ε, και και δεν είναι, αυτά, δεν είναι είδη που δεν είναι βαθιά θάλασσα, είναι άλλα είδη. Ε, είμαστε ακριβώ εδώ πέρα για να τα συζητήσουμε πώ δεν θα υπάρχουν αυτέ οι αρνητικέ παράλληλε επιπτώσει και ήδη είμαστε σε συζητήσει με συναδέλφου. Όσον αφορά απάντηση Επιτροπή, το Death Limitation δεν υπήρχε στην πρόταση τη επιτροπή. Πάλι θέλω να επαναλάβω ότι ο στόχος μας είναι να μην έχει κανένα impact, καμιά επίπτωση σε αλία άλλων ειδών από την ε, βαθιά θάλασσα. Για... Η κυρία Φράγκα είπε γιατί δεν ψαρεύουμε με τρόλες σε αμμώδες περιοχές, στις περιοχές που, έχουμε, που ξέρουμε ότι πλέον δεν υπάρχουν χωράκια και σφουγγάρια. Τα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ακόμα και εκεί πέρα που έχουμε ψαρέψει επανειλημμένα με τρόλες και έχει γίνει καταστροφή και ακόμα και εκεί πέρα που είναι αμμώδεις περιοχές βρίσκουμε θύλακες κοραϊών και σφουγγαριών. Ακόμα και σε εκείνες τις περιοχές χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τέλος, ε, θα ήθελα να κλείσω με ένα σχόλιο. Δεν είδα κάποιο συνάδελφο να... Ήταν ο κύριος Ντέιβις βέβαια επειδή υπήρξε μια επίθεση εναντίον τη κυρία Ρόσμπαχ, θέλω να θυμίσω στου αδέλφου, η κυρία Ρόσμπαχ είναι μέλο αυτή τη επιτροπή. Μπορεί να ήταν και η συγκήτρια ε, τη έκθεση στην ε, ΕΜΒ, αλλά είναι μέλο αυτή τη επιτροπή και την, ε, επειδή συνεργαζόμαστε όπω με όλου του κοιόδη συγκητέ, ε, παρακαλώ όλοι να, να θυμούνται το γεγονό ότι δεν είναι ένα εξωγήινο από κάποια άλλη επιτροπή, είναι συναδελφό μα από εδώ μέσα. Bien. Muchas, muchas... Μάλιστα, πολύ σας ευχαριστώ. Νομίζω ήδη επαρκώς συζητήσαμε αυτό το θέμα. Και έτσι λοιπόν, καθώς θα έχουμε και ευκαιρία στο μέλλον να συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Αληθεύει σε σχέση με αυτό το θέμα και με τις τροπολογίες, υπήρξε κάποια απόφαση σε σχέση με τους συντονιστέ και θα επικυρωθεί στο αντίστοιχο σημείο η απόφαση αυτή των συντονιστών. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη με την παρουσίαση παρουσίαση του σημειώματος σε σχέση με το συγκρουόμενο θέμα για τους κορμοράνους μεταξύ αλληλεία και προστασίας πτηνών. Σε σχέση με το θέμα αυτό από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου θα μας ενημερώσουν σήμερα. Έχετε αυτό το σημείωμα. Θα ακούσουμε λοιπόν σήμερα μια σύντομη παρουσίαση για αυτή την έκθεση από έναν από συντάκτες του σημειώματος, τον κύριο Γιάν Κόουτς του Εθνικού, του Εθνικού Ιδρύματος αυτού του Πανεπιστημίου από αυτή τη χώρα. Έχει τον λόγο άμεσα για να μας κάνει αυτή την παρουσίαση. Σύντομα παρακαλώ, όσο το δυνατόν περιεκτικότερα και από πλευράς όλων των Ευρωβουλευτών να υπάρχει ευκαιρία και έχουν την έκθεση και μπορούν έτσι σε μεγαλύτερο βάθος να ενημερωθούν. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή. Έχουμε ήδη, ήδη ακούσει, δεν σας κουράσω παραπάνω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ένα θέμα ακόμα, γιατί νομίζω ότι σε σχέση με τα έδρανα των Ευρωβουλευτών δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε αυτό. Σύμφωνα με τον κύριο Σάντσες Προεθέντο και μια και έχει προχωρήσει ο χρόνος, αποφασίσαμε το σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης να περάσει στην επόμενη συνεδρίασή μας. Δεν θα καλυφθεί σήμερα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Αν συμφωνείτε λοιπόν αυτό θα κάνουμε, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο ούτως ή άλλως να το συζητήσουμε σήμερα. Εντάξει λοιπόν. Ωραία, έχουν φύγει ήδη πολλοί κιόλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το 18 το διαγράφουμε από την ημερήσια διάταξη, το εξετάσουμε υστερότερα. Συνεχίστε παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ και πάλι πρόεδρε. Αυτό που σας παρουσιάσω είναι ένα πολύ αντιφατικό θέμα στην Αλία και στο θέμα της προστασίας της Αλίας και των ειδών. Είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει την Επιτροπή αρκετές φορές στο παρελθόν. Είναι η διαμάχη μεταξύ αλίας και προστασίας των ειδών και δι του κορμοράνου. Θα παρουσιάσω την έκθεση εν συντομία Και αυτό το οποίο θα καλύψω βασικά είναι πέντε τομείς. Θα αναφερθώ τηλεγραφικά στη φύση της ε, διαμάχης αυτής, ε, στην ε, κατανομή των πουλιών και την πληθώρα, τα, τα ποσοτικά στοιχεία, τις επιπτώσεις στην αλία και στις πηγές της αλίας, στις τρέχουσες ε, δράσεις για την επίλυση των επιπτώσεων, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και εν τέλει την παρουσίαση ορισμένων συστάσεων. Αυτή η, το θέμα, αυτή η διαμάχη ξεκίνησε επειδή υπάρχει ένας ε, αυξητικός ε, αριθμός κορμοράνων σε ευρωπαϊκά δάφη στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη αντίθεση μεταξύ εκείνων που θέλουν να προστατεύσουν τους κορμοράνους και εκείνων που ασχολούνται με την αλία και την ε, υδατοκαλλιέργεια, την ε, ηχθειοκαλλιέργεια. Ε, το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε ένα ψήφισμα για ένα κοινό πρόγραμμα διαχείρισης ο, ένα από τα πρώην μέλη σας, ο κύριος Κίντερμαν, είχε παρουσιάσει αυτή την πρόταση, αλλά χρειαζόταν τότε μία πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών που θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτές από τους ενδιαφερόμενους του τομέα και η Κομισιόν είχε πει τότε ότι αυτή δεν ήταν η πιο κατάλληλη λύση. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησαμε το 2008 και ας δούμε που βρισκόμαστε σήμερα. Η σημερινή κατανομή των ε, πουλιών αυτών του Κορμοράνου καλύπτει ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Δεν είναι τόσο ο ορισμός τους η πληθώρα τους, αλλά το, η εποχιακή τους μετακίνηση. Μετακινούνται, αποδημούν, ας πούμε, από τις βόρειο-ανατολικές περιοχές σε νότιο-ανατολικές περιοχές και διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ζώνες αναπαραγωγής στις χειμερινές απικίες ε, Έχουμε πολλά στοιχεία, πολλές μελέτες που έχουν γίνει για το ρυθμό αναπαραγωγής. Βλέπετε και πάλι τον χάρτη της ε, κατανομής των απικιών και το που χυμάζουν επίσης. Ε, είναι περιοχές της Βόρειας Ευρώπης αλλά και σε νότιες περιοχές της Ευρώπης. Αυτά είναι στοιχεία του Ιανουαρίου του 2003. Πολλές φορές τα στοιχεία στα οποία βασιζόμαστε ε, συλλέγονται μία φορά μόνο, άπαξ. 2006 ε, είναι τα πιο σύγχρονα, τα πιο επίκαιρα στοιχεία που έχουμε και 2003 είναι τα περισσότερα στοιχεία που έχουμε, στα οποία επενερχόμαστε συνέχεια. Πρέπει να πω ότι ε, συνεργαζόμαστε με, την, Κομισιόν και με την BirdLife International. Αν κοιτάξετε τώρα τις τάσεις της κατανομής των απικιών θα δείτε ότι ε, είναι, είναι στις παράκτιες περιοχές της ε, Βόρειας Ευρώπης και το είδος του πουλιού είναι τα σανιένσις Κορμοράνου Σαϊνένσης που είναι το πιο συνηθισμένο αναπαραγόμενο ε, η αξιοπιστία αυτού του γραφήματος ε, δεν είναι 100% εγγυημένη αλλά η τάση δείχνει ότι σαφώς ε, πληθαίνουν οι κορμοράνοι στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990 βλέπετε μια δραματική αύξηση. Υπάρχουν τώρα ποσοτικές διαφορές μεταξύ των χώρων. ή Το είδος κάρμπο είναι αρκετά ε, σταθερό, ιδίως ε, ε, πολύ μικρές αυξήσεις παρουσιάζονται στην Ορβηγία. Είναι το είδος σαϊνένσης που σας είπα που παρουσιάζει αυτά τα δραματικά αυξητικά στοιχεία τις τάσεις αυτές τις αυξητικές. Την Δανία αυξήθηκε δραματικά, συνεχεία σταθεροποιήθηκε και ο ορισμός τους και τώρα μειώνεται. Ε, πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στις ε, ενέργειες που έχουν γίνει για τον έλεγχο των πληθυσμών. Ε, έχουμε τώρα εκατομμύρια κορμοράνων στην Ευρώπη και 400 με 1000 γραμμάρια ψάρια τρώνε κάθε μέρα. Μέσω όρο 600 γραμμάρια ψαριών χρειάζεται ένα πουλί να φάει κάθε μέρα. Συνήθως τρώνε ε, μικρά ψάρια μέχρι 5-10 εκατοστά, μικρά ψαράκια δηλαδή. Α, ε, The amount of, um, Μέχρι 50 εκατοστά και πολλές φορές εάν οι κορμοράνοι είναι πάνω από 80 ή γύρω στους 80 κορμοράνους ανά εκτάριο ε, σε μια λίμνη ας πούμε μπορείτε να εξαφανίσει εντελώς τα ψάρια μέσα στην υδάτινη περιοχή αυτή. Είναι λοιπόν ε, ε, εξαιρετικά καλή αλής ψαριών. Ε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε ε, μας δυσκολεύουν. Ε, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να συλλέξουμε και να καταγράψουμε εμπειρικά στοιχεία, εμπειρικά δεδομένα. Ορισμένα μετρήσεις που έχουμε κάνει δείχνουν ότι το 20% της ετήσιας παραγωγής ψαριών στις λίμνες της Βαβαρίας εξαφανίζεται, μειώνεται κατά 20% ετήσιος και επίσης το 8,2% ε, στις πολωνικές λίμνες. Ε, επίσης, μεγάλες, μια μεγάλη βιομάζα ψαριών μετακινείται, ε, καταστρέφεται μάλλον τις μεγάλες λίμνες στο Οντάριο και στη Λίμνη Ήρη και περίπου ε, ε, υπάρχει μια 100% ε, μείωση των αλληλευμάτων σε ορισμένες περιοχές όπου υπάρχουν μικρές λίμνες αναψυχής με μικρά ψάρια κλπ. Το βασικό λοιπόν πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κάπως δραματικά στοιχεία από την συχθιοκαλλιέργεια στη Γαλλία, όπου έχουμε περιπτώσεις όπου σε ορισμένες φάρμες έχουν μειωθεί κατά 50% η ετήσια απόδοση, κατά 47% στην Κροατία και έχουμε εξετάσει και στοιχεία από τη νότιο-ανατολική, ε, από τη ΣΥΠΑ, νότιο-ανατολικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ε, η οικονομική απώλεια έχει μετρηθεί περίπου στα 25 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ε, είδε, λοιπόν όχι μόνο η απώλεια των ψαριών και η μείωση των αποθευμάτων, αλλά Υπάρχει και η συμπεριφορά των ψαριών που ε, μετατρέπεται λόγω της απειλής από τα πουλιά, προσπαθούν και φεύγουν από τα, τις προστατευόμενες περιοχές, ε, ε, πληγώνονται. Σε αυτά δεν έχουμε τόσα πολλά στατιστικά στοιχεία, αλλά επιφέρονται ζημίες, ζημίες στο σώμα των ψαριών και στη συμπεριφορά τους in Και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Επίσης υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Οι κορμοράνοι ε, επηρεάζουν τα οικοσυστήματα διότι είναι πολύ επιλεκτικά πουλιά όσον αφορά το είδος της τροφής και έτσι ε, επηρεάζουν τις δυναμικές ροές των οικοσυστημάτων, τα, δίκτυα, τα διατροφικά δίκτυα που αναψίσονται στα οικοσυστήματα, καταστρέφουν τα ορισμένα είδη, τα δάση, τα δέντρα, ε, με περιτώματα, γεμίζουν με περιτώματα το, το έδαφος και αυξάνουν την περιεκτικότητα σε αζωτούχα σουσίες. Επίσης ε, επηρεάζουν τα τσόφια από τα αυγά τους την, ε, οξύτητα των εδαφών και επίσης αφήνουν όλα τα, τα ψόφια νεογνά και αυτά είναι αρνητικά στο περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν ε, και οικολογικές ε, επιπτώσεις που αντιβαίνουν ε, τις συναφείς οδηγίες και τα μέτρα που επιβάλλουν. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν ορισμένα μέτρα. Αυτά που έχουν προταθεί διαφέρουν πάρα πολύ από την εξόντωση σε έλεγχο των, των πληθυσμών, στο να τους τρομάξουμε με κάποια μέσα, να φύγουν, να απομακρύνονται από τις ηχθειοκαλλιέργειες, να μπορούμε να, να απομονώσουμε ορισμένε περιοχές να μην πηγαίνουν εκεί και να, να μπορέσουμε να έχουμε ψάρια τα οποία ναι μεν ε, μπορούν να τα πιάσουν αλλά δεν μπορούν να πετάξουν επειδή είναι βαριά ε, διάφορα μέτρα πρέπει να τονίσω ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει στο διαδίκτυο ένα εργαλείο, ένα, μια έκθεση αυτή για τους κορμοράνους και να μπορείτε να έχετε όλη πρόσβαση. Έχουμε σκοπό να την βάλουμε στο διαδίκτυο. Τώρα, ε, εάν η εξόντωσή τους, ε, τα θανατηφόρα μέτρα είναι κατάλληλα, θα πρέπει για να γίνει αυτό να επιβληθεί μία απόκληση από το άρθρο 9 της οδηγίας για, την προστασία, για τα πτηνά. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα, μια ουσιαστική θεμελιώδης αρχή την οποία πρέπει να προσέξουμε. Από το 2001 μέχρι το 2012 250.000 κορμοράνοι έχουν θανατωθεί ε, για να αποφευθεί η σοβαρή ζημιά στη, στα ψάρια και τα, ε, τα μισά πουλιά από αυτόν τον αριθμό, δηλαδή από τις 250.000, έχουν σκοτωθεί στη Γαλλία. Το άλλο θέμα είναι ότι το άρθρο 9 και η οργάνωση Life International πιστεύει ότι το άρθρο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του πληθυσμού των κορμοράνων και για την ε, θανάτωσή τους. Υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη περιοχή, το oiling, ε, σε, σε περιοχές αναπαραγωγής, που προτείνεται, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε στοιχεία για να ξέρουμε αν το μέτρο αυτό είναι αποτελεσματικό. Εγώ πιστεύω ότι η προσπάθεια ελέγχου του πλουθυσμού τοπικά, σε τοπικό επίπεδο, δεν είναι επιτυχής, διότι αν ας πούμε εξοντώσεις ένα τοπικό πληθυσμό, ένα κοπάδι κορμοράνων, ε, μετά θα έρθει ένα άλλο να πάρει τη θέση του. Ε, τώρα, πώς μπορούμε να αποφύγουμε ε, την, ε, απώλεια των ψαριών ε, και να, τα πιάνουν οι κορμοράνιδοι, την επίθεση τους δηλαδή. Το θέμα είναι ότι ό,τι μέτρα λάβουμε προς εκφοβισμό των κορμοράνων θα εκφοβήσουν και τα ψάρια. Και, και ούτε αυτό είναι κατάλληλο. Τώρα, μεγάλες ε, ενέργειες, ενέργειες μεγάλης κλίμακας για προστασία των ξιοκαλλιεργιών, ε, με δίκτυα, κάλυψη των ε, δεξαμενών υψηλοκαλλιέργειας με δίκτυα. Αυτό θα εμποδίσει και τους διαχειριστές και το προσωπικό να δουλέψει στις μονάδες αυτές. Όπως είπαμε, μπορεί σε τοπικό επίπεδο ορισμένα από αυτά μέτρα μερικώς να είναι αποτελεσματικά, αλλά σε μεγαλύτερο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό δεν είναι. Αποζημίωση, αποζημίωση στην Τσεχία, παραδείγματο χάρη, εκεί γίνεται μεγαλύτερη ζημιά στις ηχθειοκαλλιέργειες, μονάδες ηχθειοκαλλιέργειες. Ε, πώς θα μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος της αποζημίωσης. Ε, και πολλές φορές γίνεται μια εφάπαξη καταβολή όταν γίνει η ζημιά. Ε, μέτρα διαχείρισης είναι μια άλλη δυνατότητα που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Δεν υπάρχει όμως μια ε, σύγχρονη διαχειριστική προσέγγιση και δομή σε όλες αυτές τις ε, μονάδες. Η Βόρεια, Αμερική από το Οντάριο, από τις μεγάλες λίμνες που έχουν μεγάλα συστήματα, έχουν υιοθετήσει διαχειριστικά προγράμματα μεγάλης κλίμακος που έχουν επιτύχει, ήταν αρκετά επιτυχημένα για τον περιορισμό των κορμοράνων. Ορισμένα από τα προβλήματα που έχουμε για να μπορέσουμε και να βρούμε λύσεις ε, το βλέπετε εδώ είναι ένα κλασικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης ε, κορμοράνων και ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παραδείγματο χάρη η, η, το, η, τοξικότητα στο, σε, στις οικολογικές περιοχές, η επιρροή των ε, ουσιών που μολύνουν την διατροφική αλυσίδα, η επίδραση των κορμοράνων ε, στην αλία, όλα αυτά είναι επιστημονικά θέματα, η τοξικότητα, οι μολυντές, η... Ε, αλλά βλέπετε ότι τα στοιχεία είναι αρκετά περιορισμένα που έχουμε μέχρι τώρα. Περιορισμένες πληροφορίες, περιορισμένα δεδομένα, τα οποία, πάνω στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Και ε, δεν, παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις στην αλία, δεν ξέρουμε συγκεκριμένα σε ποια είδη αλίας. Πολύ, έχουμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη παινία πληροφόρησης. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τη ζημιά που γίνεται μπορούμε να αξιολογήσουμε τη σοβαρότητα της ζημιάς, αλλά και πάλι εδώ ε, έχουμε υποκειμενικούς όρους. Πώς αξιολογούμε τη σοβαρότητα και πόσο μεγάλη είναι η ζημιά. Γενικά, όποτε προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κανονισμούς στην αλία, ε, προσπαθήσαμε να συλλέξουμε στοιχεία αν επανέκαμψε ε, η Ορισμό των ψαριών. Κάτι λίγα στοιχεία έχουμε από την Ελβετία, πολύ περιθωριακά και ελάχιστε πάλι πληροφορίε για την ανάκαμψη και για τις επιπτώσεις των μέτρων που επιβλήθηκαν. Επίσης μας ενδιαφέρει ε, πώς αντιδρούν οι, οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι αλληλείς, οι περιβαλλοντολόγοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι των ε, συναφών τομέων, όχι μόνο οι αλλοί, ε, πώς θα αντιδρούν σε αυτό το πρόβλημα. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να συλλέξουμε και τα τη, στοιχεία για την ανθρώπινη πτυχή. Εδώ βλέπετε στοιχεία από την Βασιλική Ένωση Προστασίας Πτηνών, την RSPB στο Ενωμένο Βασίλειο, στο Βασίλειο και βλέπετε εδώ ένα άρθρο ε, το οποίο παρουσιάζει τις ριζικά αντίθετε απόψεις μεταξύ των υπερμάχων των κορμοράνων και των υπερμάχων των ψαριών. Ε, ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα και γίνονται πολλές εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού όπου παρουσιάζονται ακριβώς αυτά τα άρθρα ε, και από τις δύο απόψεις, από τις δύο πλευρές έχουν εκπονηθεί ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικά προγράμματα. Υπάρχει αυτό στο Ιντερκαφέ, όπου μπορείτε πάλι να διαβάσετε τη διαμάχη και τα ε, στοιχεία της ε, συζητήσεις που έχουν γίνει μεταξύ των αντίθετων πλευρών το θέμα είναι αυτό που ρωτάω εγώ. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται με το καλύτερο τρόπο. Οι πληροφορίες αυτές και η όλη συζήτηση παρουσιάζεται συνήθως στο διαδίκτυο, αλλά οι αλληλείς που μένουν σε απομακρυσμένα μέρη είναι ενήμεροι, έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου από το 2008 η έκθεση του κυρίου Κίντεμαν, το ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Κοινό Διαχειριστικό Πρόγραμμα αλλά όπως σας είπα τότε η Κομισιόν δεν το υποστήριξε οι, δι, οι διαφορές αυτές που υπάρχουν είναι εξαιρετικά έντονες, εξαιρετικά δυναμικές εμπλέκονται κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές ε, πτυχές δεν είναι μόνο το, το πουλί τρώει τα ψάρια και πρέπει να προστατέψουμε το ψάρι. Εδώ έχουμε πολλές άλλες περίπλοκες ε, πτυχές και επίπεδα στα οποία πρέπει να εμβαθύνουμε. Ε, όπως σας είπα λοιπόν πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις στην κοινωνία, τις επιπτώσεις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις οικολογικές επιπτώσεις. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Αυτό έχει λεχθεί πολλές φορές στο παρελθόν και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Μπορούμε μόνο να, μπορούμε να προχωρήσουμε με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. πρέπει λοιπόν καταρχάς να βελτιώσουμε την, ε, τα στοιχεία που έχουμε, τα, τα επιχειρήματά μας, να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε ε, και να καταλάβουμε και να αναλύσουμε επιστημονικά τους λόγους για, την, για τους οποίους οι κορμοράνοι διευρύνουν τις περιοχές και την παρουσία τους στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να διευρύνουμε την, τις γνώσεις μας για την συμπεριφορά των πουλιών, πού αναπαραγάγουν, πού τρέφονται, με, τι τρέφονται. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρουν οικονομικές και κοινωνικές πλευρές του ζητήματος ε, και μόνο αν έχουμε αυτά τα στοιχεία μπορούμε να προχωρήσουμε στην λήψη αποφάσεων. Μπορούμε να αποτανθούμε στην Αυστραλία, στην Αμερική, εκεί που υπάρχουν περισσότερα στοιχεία αντί να βασιζόμαστε μόνο σε αυτές τις ριζικαία αντίθετες, πολλωμένες και φορτισμένες απόψεις της μιας ή της άλλης πλευράς. Πολύ πιο περίπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα εμπλέκονται σε όλο αυτό το ζήτημα. Θα επανέλθω λοιπόν στις δυνατότητες της διαχείρισης, της στρατηγικής διαχείρισης, χρησιμοποιώντας το αμερικανικό παράδειγμα έχουν έξι εναλλακτικέ λύσεις και έχουν και τη στρατηγική για να λύσουν το πρόβλημα. Έχουν εξετάσει τα συγκεκριμένα θέματα, έχουν εξετάσει τις απαντήσεις σε έξι διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι καμία παρέμβαση. Το δεύτερο ήταν να προσπαθήσουν να φοβήσουν τα πουλιά χωρίς να τα πυροβολήσουν. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα θα πάει κάπου αλλού. Ε, τρίτον, περιορισμός τοπικά της ε, ζημιάς ε, σε συγκεκριμένες αλλιευτικές περιοχές. Μετά περνάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, παρακολούθηση προσεκτική των, του αριθμού των πτηνών και τέλος περιφερειακή προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού των πτηνών και τελευταία, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα είναι ένα ελεύθερο κυνήγι. Νομίζω ότι αυτό είναι το υψηλότερο σε κλίμακα στο οποίο μπορεί να φτάσει κανείς πλήρης απελευθέρωση του κυνηγίου των κορμοράνων. Το θέμα εδώ θέτει κάποια προβλήματα δεοντολογίας σε σχέση με την διατήρηση του είδους. Τέτοιου είδους ε, μεγάλης κλίμακας μειώσεις του πληθυσμού των πτηνών δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Υπάρχει αυτό το οποίο γίνεται στη Δανία, το λεγόμενο oiling, αλλά αυτό δεν ξέρω αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την κοινωνική διάσταση με την περιβαλλοντική διάσταση. Υπάρχουν οι κορμοράνοι, υπάρχουν τα λόμπι υπέρ των κορμοράνων, υπάρχουν τα λόμπι για την αλληλεία και τη διατήρηση της οικονομικής αυτής δραστηριότητας. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ε, σε κάθε τομέα τι έχει σημασία. θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και να πείσουμε γιατί πρέπει να ρυθμίσουμε τους πληθυσμούς των κορμοράνων και θα πρέπει επίσης να συνδυάσουμε τις λύσεις και όχι να ακολουθήσουμε αποκλειστικά μία πορεία. Να βελτιώσουμε λοιπόν τις ε, συνθήκες Υπάρχουν οι δυνατότητες να προχωρήσουμε σε επιβολή μίας λύσης, αυτό όμως απαιτεί ίσως ε, κάποιες αλλαγές σε επίπεδο κεντρικού συντονισμού, σε επίπεδο θεσμικού συντονισμού. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή η οποία συγκεντρωτικά να προσπαθεί να ελέγξει τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν στους πληθυσμούς Οι κορμοράνοι δεν θα εξαφανιστούν πάντως, δεν υπάρχει τρόπος για να εξαφανιστούν πλήρως. Οι κορμοράνοι είναι εδώ και θα παραμείνουν εδώ. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μια προσπάθεια βελτίωσης ε, των τρόπων ε, μεταχείρισης αυτού του ε, πτηνού. Απαιτούνται μελέτες και θα πρέπει ίσως να ξεφύγουμε από κάποιους περιοριστικούς δείκτες όπως η τοξικότητα και η μείωση της τροφής και να περάσουμε σε ευρύτερες μελέτες οι οποίες ε, να μας δίνουν την δυνατότητα να ελέγξουμε το πρόβλημα καλύτερα. μέσω συντονισμού, μέσω μιας κάποιας κεντρικής αν θέλετε υπηρεσίας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε.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 Llevan dos días diciéndolo y Θα προσπαθήσουμε την άλλη φορά να βελτιώσουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε τίποτα. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν καθηγητά για την παρουσίασή σας. Εμπεριέχονται πολλά σημαντικά στοιχεία καταδεικνύουν μια δραματική ανάπτυξη όσον αφορά αυτά τα ηχθιοφάγα πτηνά και τις απώλειες που υπάρχουν όσον αφορά ηχθειοκαλλιέργειες πράγμα το οποίο δημιούργησε σημαντικές τριβές μεταξύ περιβαλλοντολόγων, προστα... Ε, υπερμάχων της προστασίας του περιβάλλοντος και αλλιέων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία και μόνη βέλτιστη μέθοδος ε, δράσης. Διάφορες μέθοδοι πρέπει να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουμε αυτά τα πράγματα, αυτή την κατάσταση και με συντονισμό σε διεθνές επίπεδο αυτών των δράσεων θα είμαστε οι πιο αποτελεσματικοί στη δράση μας. Κάνω λόγο για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο πρόγραμμα διαχείρισης και τη σύσταση για ένα τέτοιο πρόγραμμα ώστε να μειωθούν οι απώλειες που προκαλούνται από τους κορμοράνους στην Αλία και στην, ε, ε, στις Υπό αυτό το πρίσμα η παρουσίαση που έγινε είναι ιδιαίτερα αξιόλογη διότι συμπεριλαμβάνει πάσης φύσεως στοιχεία και καταδεικνύει ότι υπάρχουν και διαφορές μεταξύ απόψεων επιστημόνων. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει ε, θετική επίπτωση, άλλη αρνητική. Αυτό το παράδοξο όμως αυτό το επίμαχο θέμα μπορεί να επεξηγηθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, οι κορμοράνοι ως ηχθειοφάγα πτηνά μπορούν να διαδραματίσουν και κάποιο θετικό ρόλο. Όχι όμως σίγουρα όταν είναι υπερβολικός ο αριθμός τους και όταν επεκτείνονται σε άλλες περιφέρειες και ζώνες ε, και παρισφρέουν και δρούν με καταστροφικό τρόπο εκεί. επιπλέον, σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις στις υδατοκαλλιέργειες και στο εισόδημα των ε, όσων εκμεταλλεύονται αυτές και των αλλιέων. Επίσης, μια πανευρωπαϊκή στρατηγική σε σχέση με αυτό το στόχο επισημαίνεται ότι είναι ανάγκη να έχουμε ακριβώς μια πανευρωπαϊκή στρατηγική που θα λειτουργήσει. Εγώ πιστεύω ότι η αποτυχία των περιφερειακών στρατηγικών ως μέθοδος προσέγγιση απορρέει από την απουσία μιας τέτοιας πανευρωπαϊκής, πανενοσιακής προσπάθειας. Και βλέπουμε εδώ ότι μειώνονται διαρκώς τα αλλιεύματα ενώ ο αριθμός των κορμοράνων αυξάνεται και η αρνητική τους επίπτωση και αυτή αυξάνεται. Γι' αυτό δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια και απλά ως παρατηρητές ε, να παρακολουθούμε ουδέτερα αδρανώς το τι συμβαίνει. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να δράσουμε, μια και είναι ιδιαίτερα επιθετική η κορμοράνη και παρισφραίουν με τέτοιο τρόπο με την αύξηση σε αριθμούς τους ε, με τρόπο αρνητικό. Φυσικά είναι, θετικό, είναι σαφές ότι με συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την ε, υποστήριξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Αλία και το Διατοκαλλιέργειες θα είναι η πιο εύθετη λύση που θα μπορούσε να υιοθετηθεί. Ιδιαίτερα όταν γίνεται αυτή η πρωτοβουλία, αναλαμβάνεται η πρωτοβουλία υιοθέτηση μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής όπως είναι αναγκαία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο καθηγητή Κότς για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του όπου πιστεύω και πρέπει να το πω ότι κάποιοι βασικοί κανόνες που υπάρχουν στην ίδια τη φύση δεν πρέπει υποχρεωτικά επιστημονικά να αναλύονται ένα τέτοιο πτηνό το οποίο βρίσκεται πάνω πάνω στην αλυσίδα και που ε, καταλήγει σε αυτούς τους αριθμούς ε, στους οποίους καταλήγουμε με τους κορμοράνους είναι απλή κατάσταση. Ας μην εκπλησώμεθα, ίσα ίσα παίρνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό είναι αναγκαίο για τέτοιου είδους μεταναστευτικά πτηνά ε, να ε, σχεδιάσουμε μια παρέμβαση ευρωπαϊκή για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Το Κοινοβούλιο έχει πλήρως τοποθετηθεί από αυτόν, το είπατε καθηγητά, το 2008 ελήφθη η απόφαση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό δεν έλαβε δράση. Σχετικά ελάχιστα έκανε το νομοθέτημα για την προστασία της ορνηθοπανίδας και την προστασία των βιοτόπων και η οδηγία για την... Στο εδάφιο 9, το αναφέρατε σωστά, το επιτρέπει να γίνει αυτό. Αν ένα συγκεκριμένο είδος έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα είδη, τα οποία εξοντώνει, ε, τότε μπορεί άμεσα να υπάρξει άμεση επέμβαση ή παρέμβαση. Και περί αυτού πρόκειται ακριβώς εδώ άμεσα. Τι γίνεται, για παράδειγμα, με την προστασία του ευρωπαϊκού χελιού. Βρίσκεται βρίσκεται στον κόκκινο κατάλογο επαπειλούμενων ειδών και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία το ίδιο ισχύει. Μόνο πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να τους προστατέψουμε. Και έχουμε και μία εικόνα, μία φωτογραφία με ένα κορμοράνο που στο ράμφος του έχει ένα χέλι. Τι είναι αυτό, σύμβολο προστασίας του περιβάλλοντος. Ας συζητήσουμε σοβαρά σε βάθος πώς θέλουμε να προστατέψουμε αυτά τα είδη. Εκεί όπου υπάρχουν οι ζημιές που γίνονται στις παράκτιες περιοχές ε, πρέπει κάτι να, να κάνουμε και να δράσουμε. Όπως είπατε κύριε καθηγητά πρέπει με όλους τους εμπλεκόμενους να καθίσουμε γύρω από μια στρογγυλή τράπεζα και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε, να αναχαιτήσουμε αυτό το φαινόμενο. Οι κορμοράνοι διεισδύουν όλο και περισσότερο στην ενδοχώρα. Περνάνε και σε μικρά ποτάμια και λίμνες στο εσωτερικό, στα Μεσόγεια. κάτι να γίνει αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των κορμοράνων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, για παράδειγμα, και της γονιμότητας ή του πολλαπλασιασμού των ε, κορμοράνων, ώστε να μην πολλαπλασιάζονται έτσι. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική ρύθμιση γεννήσεων ή τέλο πάντων του πολλαπλασιασμού των κορμοράνων. Αυτή είναι η πρότασή μου. Υπάρχουν πολλά επιστημονικά πορίσματα και στη Γερμανία. Το Πανεπιστήμιο Ρόστοκ πήρε εντολή και από την περιφερειακή κυβέρνηση της Πομερανίας, ε, δυτικής Πομερανίας με υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Έχουμε πλημμυρίδα, κατακλυσμό κορμοράνων και αυτό το οποίο έχουν επίπτωση μεγάλες απώλειες ψαριών, αν υπολογίσετε χιλιάδες κορμοράνοι επί χι ε, βάρος ε, ηχθείων, αυτό τι κάνει. Τόνους ολόκληρους ε, ηθείων ε, ε, που εξοντώνονται. Είχα πάει στον ποταμό Έλβα και εδώ πραγματικά όσον αφορά τους τόμου, τους, ε, τις περιοχές όπου αφήνουν τα αυγά τους ε, πολλοί πληθυσμοί ε, αλλιευμάτων που εξοντώνονται πρέπει να προστατέψουμε αυτά τα είδη. Είναι ένα θέμα που πρέπει σε βάθος και σοβαρά να το λάβουμε υπόψη. Όχι μόνο για να μην υπάρχει ζημιά στην αλία αλλά εδώ πρόκειται για εξόντωση ολόκληρων ειδών. Σε δύο λεπτά, λιγότερο από δύο λεπτά ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Συνδέεται με αυτό με το ότι τελειώσαμε χθε δυόμιση ώρε νωρίτερα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τι ώρε αυτέ καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα των κορμοράνων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα Συμφωνώ και με τον κύριο Κούν και με τον κύριο Βαλένσα ότι θα πρέπει να το επανεξετάσουμε προσεκτικά και με την σωστή μεθοδολογία. Έχουν υπάρξει ορισμένες καλές πρωτοβουλίες Έχουμε τη λεγόμενη εργαλειοθήκη η οποία είναι διαθέσιμη και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και η UNEP στα τέλη της δεκαετίας του 90 υιοθέτησε ένα πρωτόκολλο σχετικά με τη μείωση των πληθυσμών των αρπακτικών. Υπάρχει δηλαδή ένα πρωτόκολλο εγκεκριμένο από τα Ηνωμένα Έθνη που επιτρέπει να δει κανείς τις συνέπειες ε, της, ε, ε, της θανάτωσης τμήματος των ζώων. Επί τη βάση λοιπόν όλων αυτών νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση, να θέσουμε ερωτήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την πρόοδο που έχει υπάρξει σχετικά με το πρόγραμμα δράσης ΣΥΜΠΕΛ δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το κάνουμε τώρα πια. Και να θέσω στον εμπειρογνώμονα μία συγκεκριμένη ερώτηση. Είδαμε περιέργεια ότι οι κορμοράνοι αυξήθηκαν παντού, αλλά όχι στην Ορβηγία. Στην Ορβηγία υπήρξε μία συνεχής αντιμετώπιση, προσπάθεια μείωσης του είδους και στην Ορβηγία γνωρίζουμε επίσης και το ζηλεύουμε έχουν πάρα πολύ ψηλά επίπεδα αλλιευμάτων επίσης. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε αυτό. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο καθηγητής ώστε να απαντήσει σύντομα σε αυτές τις ερωτήσεις. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επανέρχομαι στο ερώτημα για την Νορβηγία. Καταρχάς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για τα στοιχεία που παρουσίασα υπάρχουν να τα οποία πληρώθηκαν ε, μετά από διάφορες ε, μελέτες που έγιναν από πηγές που δεν είναι και τόσο αξιόπιστες. Άρα λοιπόν με μεγάλη επιφυλακτικότητα εξετάζουμε τα στοιχεία αυτά. Και ενδέχεται οι πληροφορίες που έχουμε και τα στοιχεία της Νορβηγίας να μην είναι 100% ακριβή. Το άλλο θέμα είναι ότι στην Νορβηγία επικρατεί το είδος του κορμοράνου κάρμπο, το οποίο όπως σας είπα δεν είναι τόσο... Ε, δεν, δεν εμφανίζεται τόσο πολύ στις άλλες περιοχές και είναι συνήθως στις παράκτητες περιοχές, σε λίμνες και εμφανίζει ένα σταθερό πληθυσμό. Ο, ο του είδους κάρμπο δεν αυξάνεται τόσο πολύ όσο ο άλλος πληθυσμός του είδους συνένζης όπου εμφανίζεται, εμφανίζεται δραματική αύξηση όπως είδατε. Και επανέρχομαι σε κάτι άλλο που είπαν. Οι προλαλήσαντες είναι τα εάν τα, οι μελέτες αυτές βασίζονται σε αξιόπιστες πηγές και στοιχεία. Ε, εδώ πάλι έχουμε ελλείψεις. Όταν θέλουμε να συλλέξουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις αναλύσουμε, πρέπει να εξετάσουμε όλες τις προοπτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, περιβαλλοντικές ε, ενώ παλαιότερα είχαμε μία μοναδική ή ενιαία πηγή ε, πληροφόρηση, συλλογής πληροφοριών. Ε, χρησιμοποιούσαμε παραδείγματο χάρη στοιχεία ιατρικά, ενώ τώρα χρησιμοποιούμε μία ποικιλομορφία δεδομένων. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Διάφορα δεν υπάρχουν τίποτα στα διάφορα και η προαναγγέλω για τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές. Έχουν αποσταλεί σε εσά, έχετε το έγγραφο και αν έχετε κάποια παρέμβαση παρακαλώ. Η ημερομηνία επόμενης συνεδρίασης Βρυξέλλες 22 Απριλίου το απόγευμα. 23 το πρωί από το απόγευμα και το, το πρωί και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.